Okay, good morning. Let's start our work today. Καλημέρα σας. Αρχίζουμε. Σχέδιο μέσα διάταξης. Έχετε καμία πρόταση, κανένα σχόλιο, όχι. Τότε θεωρώ εγκεκριμένη την ημερήσια διάταξη. Ε, επιτρέψτε μου να σας κάνω μερικές ανακοινώσεις εξ ονόματος της Προέδρου μας. Στις 26 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή μας συνεδριάζει μαζί με εθνικούς βουλευτές που έχουμε προσκαλέσει στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της έκθεσης του κυρίου Γκοζές. Για να συμμετάσχετε στην απογευματινή συνεδρίαση πρέπει να σας πω ότι θα αρχίσει ακριβώς στις 3 να το γνωρίζετε. Μετά την ανταλλαγή αυτή απόψεων θα ψηφίσουμε αμέσως. για το σχετικό θέμα που έχουμε να ψηφίσουμε για τις ε, πληρωμές με κάρτα μέσω του διαδικτύου και μέσω κινητών τηλεφώνων. Για το τριμερή διάλογο έχουν γίνει κάποιες πρόοδοι με τον κύριο Γοζές Και επίση θα συζητηθεί το θέμα των κρατών που χρειάζεται βοήθεια και με ποιο τρόπο θα τη ζητούν. Η επόμενη συνεδρίαση ε, τριμερίου διαλόγου ε, θα αφορά την λέξη της κυρίας και θα γίνει στις 4 Οκτωβρίου. Πριν αρχίσουμε τη συζήτηση πρέπει να σας κάνω και άλλη ανακοίνωση. Μια πρόταση ε, για την Τραπεζική Ένωση και σχετική ακρόαση ε, σε συνεργασία με τους συντονιστές και τους ε, εισηγητές μετά την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε την περασμένη εβδομάδα ζήτησε η Γραμματεία να διοργανωθεί η έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής την Τετάρτη 10η Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι 9 με 1 για να διεξαχθούν ακροάσεις για την εξής νομοθετική πρόταση, Τραπεζική Ένωση και Διαχείριση της Κρίσης. Τώρα, για σήμερα το πρωί έχουμε δύο σχετικές μεταξύ τους εκθέσεις, την έκθεση κυρία Τάισεν και την έκθεση του κυρίου Γκίγκολτ προτείναμε να γίνει κοινή συζήτηση. Είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και για τις δύο Και θα δώσω το λόγο στην κυρία Τάισεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, Υποθέτω ότι οι παρόντες συνάδελφοι στη συνεδρίαση που αφορά αυτές τις δύο προτάσεις γνωρίζουν, διάβασαν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οπότε δεν χρειάζεται να επεκταθώ ούτε να χάσουμε χρόνο στην εξήγηση. 28 άρθρα είναι αν πρέπει να τα διαβάσετε ακόμα αλλά είναι πάρα πολύ πυκνά και πάρα πολύ ε, ευρύ εφαρμογή τους. Αντάλλαξαμε απόψεις και με τον συνάδελφο Γκίγκολτ, είχαμε και μια κοινή ανάλυση, αλλά τώρα ίσως να αρχίσω με ερωτήσεις. Συμφωνείτε ως εισηγήτρια να επικεντρωθώ σε έξι σημεία για την εκπόνηση μιας έκθεσης, ε, σχεδίου δηλαδή. Πρώτον, Το θέμα των 100 εκατομμυρίων. Δηλαδή ερώτηση των 100 εκατομμυρίων. Ε, θέλουμε ένα ευρωπαϊκό μηχανισμό εποπτείας για το χρηματοπιστωτικό τομέα. Ε, θα πρέπει να αναρωτηθούμε και να απαντήσουμε γιατί εδώ και χρόνια εμείς ζητούμε μια τέτοια εποπτική αρχή και μάλιστα έχουμε διαμαρτυρηθεί και καταγγείλει το γεγονός ότι δεν έχει δημιουργηθεί νωρίτερα και η ιδέα ενός νέου μηχανισμού ρύθμισης είναι κάτι που μας βρίσκει ε, σύμφωνος. Δεύτερον, θα πρέπει ο μηχανισμός αυτός να είναι ποιοτικός, στοχευμένος και αποτελεσματικός. Τρίτον, σημείο φετήριας, μηχανισμός εποπτείας που να... Ε, συνεργάζεται καλά με την εσωτερική αγορά και να εξασφαλίζει τη λειτουργία της. Τέταρτο. Αυτός ο μηχανισμός ε, θα εποπτεύει κατά προτίμηση επιστοτικά ιδρύματα από όλη την Ένωση. Πέμπτον, να έχουμε ένα σαφή καταμερισμό ε, αρμοδιοτήτων και προσωπικών ευθυνών μέσα σε αυτό το σύστημα ε, του Ευρωπαίου Επόπτη σε σχέση με τους εθνικούς φορείς και έκτον, θα πρέπει να υπάρχει σωστή λογοδοσία. Δηλαδή, θεωρούμε ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φροντίσουμε όταν εκχωρούνται τέτοιες εξουσίες εποπτείας από εθνικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο να είναι οργανωμένη και η λογοδοσία και η ευθύνη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι δεν είναι εκεί που ασκούνται και αυτές οι εξουσίες. Και ένα τελευταίο η θέση σε ισχύ του μηχανισμού αυτού. Θα πρέπει να προσέξουμε πολύ τις ημερομηνίε και να πούμε ότι, προτείνω τουλάχιστον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το υψηλό επίπεδο της εποπτείας που απαιτείται και θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει δυνατότητα απορρόφησης από το μηχανισμό αυτό όλων των εξουσιών που του αναλογούν και επίσης να υπάρχει ένα σωστό ε, ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο για να μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει και να τεθεί σε ισχύ αυτό το σύστημα. Αυτό λοιπόν τα έξι σημεία σας προτείνω ως αφετηρία και θα παρακαλούσα να μου πείτε την απόψη σας σίγουρα οι σκιώδες ηγητές αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Εκινώντας λοιπόν από αυτή την αφετηρία πρέπει να σας πω και τα προβλήματα που με απασχολούν και με ανησυχούν. Δηλαδή, και πού χρειάζεται να δουλέψουμε και να αλλάξουμε την πρόταση. Θα πρέπει να τροποποιήσουμε κάποιες προτάσεις που λένε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε μια εποπτική αρχή ε, που ε, σε πρώτη φάση αφορά τα χρηματοπιστωτικά ε, ιδρύματα που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται στην Ευρωζώνη και ε, ε, απέναντι στην ενιαία αγορά πώς λειτουργεί αυτό. Δηλαδή έχουμε αυτό το διώνυμο 17-27. Ε, θα πρέπει να δούμε οι επιχειρησιακές εξουσίες και αρμοδιότητες πώς κατανέμονται ανάμεσα στον Ευρωπαίο ρυθμιστή και τον Εθνικό ρυθμιστή ή επόπτη. Αυτό το έχουν αφήσει στα χέρια του Ευρωπαίου επόπτη να το αποφασίζει πώς θα γίνει, με ποιο τρόπο και πότε. Όχι. Εμείς θα πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό ανάλογα με το είδος ε, του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, γιατί μπορεί κάποιο ίδρυμα να ε, ενταχθεί ε, απευθείας στον Ευρωπαίο επόπτη ή να είναι η τελική αρχή στην οποία θα απευθύνεται αφού πρώτα έχει περάσει από την εθνική αντίστοιχη εποπτική αρχή. Λοιπόν, θα πρέπει να το δούμε αυτό. Τι καθήκον θα αναλάβει κάθε αρχή και με τι θα την επιφορτήσουμε. Και για κάθε τράπεζα ε, να υπάρξει ένα βέβαια σύστημα, αλλά με συγκεκριμένο καθορισμό αρμοδιοτήτων. Επίσης, θα πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξουμε και τον τρόπο λειτουργίας αυτού του εποπτικού μηχανισμού. Δηλαδή, να κοιτάξουμε πολύ καλά το διαχωρισμό ε, της νομισματικής εντολής με την εποπτική εντολή. Γιατί ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ως κύριο λόγο να, και ρόλο να προσέχει τα νομισματικά και να ασχολείται με αυτά στην Ένωση. Λοιπόν, ο μηχανισμός εποπτείας θα πρέπει να ε, έχει αρκετά εχέγγυα για να λειτουργεί σωστά, να είναι μια καλή τραπεζική εποπτεία που να οδηγεί τελικά σε νομισματική σταθερότητα. Και αυτό μας ενδιαφέρει, γι' αυτό ε, είναι και το επιχείρημα γιατί έχει ενταχθεί αυτό στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλλά να είναι δύο διακριτές αυτές ε, οι Γιατί αν πάει κάτι στραβά με την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή ε, Τραπεζών δεν θα πρέπει να την πληρώσει η Κεντρική Τράπεζα. Μετά, ε, το Εποπτικό Συμβούλιο. Ποιο, είναι αυτός ο οργανισμός ε, που στην πράξη θα ασκεί αυτή την εξουσία. Πώς εντάσσεται αυτό στη δομή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δηλαδή, Είπαμε ότι θέλουμε όσο γίνεται περισσότερα κράτη-μέλη να συμμετέχουν. Άρα θεωρούμε ότι χρειάζονται κάποιες αλλαγές ε, από το Εποπτικό Συμβούλιο αυτό μετά. Ε, Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, EBA και η έκθεση Giggold. Ό,τι λέμε στη μία έκθεση θα πρέπει να συνάδει με αυτά που αναφέρει η άλλη έκθεση. Ε, Δηλαδή, πώς θα υπάρχει η σχέση με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή που ε, δουλεύει ανεξάρτητα, έχει καθήκοντα και εξουσίες και πώς ε, θα λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις. Και επίσης θα πρέπει να αγγίψουμε και στον τρόπο με τον οποίο ε, το Εποπτικό Συμβούλιο που θα δημιουργηθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ώστε να λαμβάνει τις αποφάσεις. Αυτά είναι τα οργανωτικά και η λειτουργία του μηχανισμού και ε, ακόμα ένα θέμα ε, είναι η λογοδοσία, σε ποιον είναι υπόλογο αυτό το όργανο και σε ποιον αναφέρεται. Είναι πολύ σημαντικό, δεν χρειάζεται να σας το εξηγήσω. Ε, θα περίμενα τις προτάσεις σας σχέση με τους άλλους πυλώνες της Τραπεζικής Ένωσης. για την εκαθάριση των τραπεζών, για τις εγγυήσει των καταθέσεων και όλα αυτά θα πρέπει να μας απασχολήσουν πώς συνδέονται μεταξύ τους και ενδεχομένω να επηρεάζει η κατάσταση των πραγμάτων σε αυτά τα θέματα και το ρόλο της επιλογής θέσης ισχύς του μηχανισμού αυτού και της εποπτείας. Λοιπόν, όπως μπορέσατε όλοι να διαβάσετε στην πρόταση κανονισμού, προτείνεται ο μηχανισμός αυτός να τεθεί σε ισχύ την 1η Πρώτου του 2013, δηλαδή σε τρεις μήνες να είναι λειτουργικός ο μηχανισμός και επιχειρησιακός. Ακούγονται διάφορα ε, και ε, υπόθηκαν και διάφορα στη Λευκοσία στη συνεδρίαση του ΕΚΟΦΗΝ. Ε, διαβάζουμε και δημοσιεύματα στον τύπο για το τι δηλώνουν άλλοι φορείς. Ο κύριος Σούλτς, πρόεδρος του Κοινοβουλίου μας, από ό,τι φαίνεται έχει κάνει και ίδιους δηλώσεις και τις διάβασα στη Frankfurter Allgemeine. Ε, κάπου θα πρέπει να ε, συζητήσουμε αν στηρίζουμε αυτή την ημερομηνία ως Κοινοβούλιο γιατί έχει και επιπτώσεις και συνέπειες ό,τι αφορά τη λειτουργία και την οργάνωση της δικής μας ε, εργασίας. Ένα τελευταίο. Θα πρέπει επίσης να κοιτάξουμε πάρα πολύ καλά ε, για την επιλογή του Προέδρου. Στην πρόταση ε, η αποπτία ε, ε, ε, έχει ως νομική βάση το άρθρο 127.6. Είχαμε κάνει μια προφορική ερώτηση στην τελευταία ολομέλεια, το ψήφισμα Μπόλ, αν θυμάστε, και πιέζαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι δύο κανονισμοί για την προσαρμογή ε, της τραπεζικής αρχής και ε, τούτοι εδώ ε, να ενταχθούν στο ίδιο πακέτο και να είναι στην απόφαση. Αλλά θα πρέπει να αλλάξει νομική βάση, γιατί αν διατηρηθεί αυτή το 167-6 ε, εντάσσεται αμέσω στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό μπορεί να έχει και πλεονεκτήματα, μπορεί να έχει και προστιθέμενη αξία για την νομισματική σταθερότητα, που είναι υπόθεση της ΕΚΤ, έχει και πολύ μεγάλη εμπειρία ε, έχει διατηρήσει και το ειδικό βάρος και το ηθικό της κύρος ε, παρά την κρίση και αυτό δεν είναι ίσονο σημασία γιατί για να επανέλθει η εμπιστοσύνη και των αγορών και των πολιτών ε, στο σύστημα είναι καθοριστικό. Ο μηχανισμός όμως εποπτείας έχει το εξή πλεονέκτημα. Αν μπει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, υπάρχει μια εφιστάμενη δομή, δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο. Οπότε λειτουργεί και γρηγορότερα και αποτελεσματικότητα από το να στηθεί από την αρχή, από το μηδέν, ε, καινούρια δομή, ένα νέο ίδρυμα, ένα νέο οργανισμό. Και επίση υπέρ τη Κεντρική Τράπεζα συνηγορεί και το γεγονό ε, ότι και το Συμβούλιο. Ε, ε, υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία και είδαμε και στα σημερινά δημοψιεύματα ότι πολλά κράτη συμφωνούν στο Συμβούλιο να ανατεθεί αυτός ο ρόλος στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει ε, ε, λόγος να κάνουμε άλλη πρόταση. Εμείς είμαστε μεν συνομοθέτης, αλλά όχι αποκλειστικός νομοθέτης. Οπότε πρέπει να σκεφτούμε τι λένε και άλλοι και ότι η ευρεία πλειοψηφία του Συμβουλίου είναι προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτά, Πρόεδρε. Ε, η ταχύτητα είναι σημαντικό. Εντάξει, μια σχετική ταχύτητα πρέπει να γίνει ε, κάποια πρόοδος. Γιατί το τονίζω τόσο πολύ. Ε, διότι η κρίση δεν έχει περάσει και γνωρίζουμε ότι και στην Ευρωζώνη, στο Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωζώνης υπάρχει πολιτική συμφωνία για τη δημιουργία ενός τέτοιου μηχανισμού εποπτείας και ότι αυτό είναι αναγκαία προϋπόθεση για να συμφωνήσουν για το μηχανισμό σταθερότητας, να ε, δίδονται άμεσα σε τράπεζες ε, χρηματικές ενισχύσεις. για να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος μεταξύ ε, των δημοσίων οικονομικών και των τραπεζικών προβλημάτων. Λοιπόν, οι καιροί δεν είναι συνηθισμένοι, είναι ακόμα κρίση. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι χρειάζεται κάποια επιτάχυνση. Μπορεί αυτά να μας δεσμεύουν περισσότερο, αλλά θα πρέπει να βρίσκουμε πάντα τις καλύτερες δυνατές λύσεις και μεγαλύτερη προκλήση είναι, πρόκληση είναι να συμβάλλουμε στην ε, επαναφορά ή την επάνωδο της εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ως εισηγήτρια πρέπει να σας πω ότι μελέτησα πάρα πολύ προσεκτικά και σε μεγάλο βάθος την ε, πρόταση, που είναι και ο ρόλος μου άλλωστε ως συγγήτρες. Υπάρχουν κάποιες ε, δυσκολίες, κάποιοι περιορισμοί και για την ε, λογοδοσία και για την εξίσωση των κρατών μελών, αν ενταχθεί αυτό το σύστημα στην Κεντρική Τράπεζα, αλλά υπάρχει περιθώριο και στο καταστατικό της και στον τρόπο λειτουργία. Δηλαδή, για να βελτιώσουμε την πρόταση και πολύ μπορούμε να κάνουμε τροπολογίες, αλλά δεν ξέρω μήπως χρειαστεί ε, να θεωρήσει το συνθήκον ε, έτσι, μακροπρόθεσμα, αλλά δεν είναι του παρόντος γιατί θα μας καθυστερήσει πολύ. Αυτά. Νομίζω ότι σχεδιαγράφησα λίγο το πλαίσιο των προβλημάτων σας είπα τα έξι σημεία από τα οποία εκείνο. Σας είπα τις ανησυχίες και τα προβλήματα που έχουμε με την πρόταση που έχει κατατεθεί. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε τροπολογίες και να ακούσω και τις προτάσεις με χαρά των συναδέλφων. Και το τρίτο είναι η επιλογή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και για την νομική βάση. Θα γίνει συζήτηση. Προσπάθησα να σας ε, αναφέρω ε, τα πλεονεκτήματα γνωρίζοντας ότι υπάρχουν και περιορισμοί πάντα. Ε, στο μεταξύ Γνωρίζουν οι συνάδελφοι ε, πώς λειτουργώ ως εισηγήτρια. Προσπαθώ πάντα να ε, έχω συμβαστικό πνεύμα για πλειοψηφία στην Επιτροπή και γενικότερα. Και για να ακούγεται η φωνή μας ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχουμε ευρία υποστήριξη στις εκθέσεις μας. Ευχαριστώ και με χαρά να ακούσω τους άλλους συναδέλφους. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. σας ε, μιας και έχουμε δύο εκθέσεις οι οποίες είναι πολύ ε, κοντά η μία στην άλλη δίνω το λόγο στον κύριο Γκίγκολντ Ευχαριστώ. Είναι κομβικό αυτό το σύστημα και το θέμα διακομματικά ε, συζητήσαμε και διαπραγματευτήκαμε για το πακέτο της εποπτείας εδώ και καιρό ήταν μακρά η διαδικασία και μεγάλη ενότητα ε, του Κοινοβουλίου από τη μια και από την άλλη ήταν ενοχλητική συμπεριφορά ορισμένων μελών του Συμβουλίου. Το αποτέλεσμα ήταν κάτι που μας γέμισε όλους με περηφάνεια, γιατί είμαστε στο δρόμο μιας ευρωπαϊκής εποπτείας ε, της χρηματαγοράς, αλλά πάρα πολύ γρήγορα φάνηκε ότι και αυτό το οικοδόμημα έχει ε, σύνορα. Κάναμε μια ακρόαση την περασμένη εβδομάδα με τους τρεις επικεφαλείς των εποπτικών αρχών και πάντα ε, τόνιζαν ότι αυτή η διπλή δομή, ευρωπαϊκή και ε, εθνική ταυτόχρονα, έχει περιορισμούς και για τους φορολογουμένους είναι και η πιο ακριβή λύση. Στις ε, δοκιμασίες αντοχής, στα stress test, τα στοιχεία που προέκυψαν ε, ξεπεράστηκαν πάρα πολύ γρήγορα από την πραγματικότητα. Και γι' αυτό περιμένουν οι πολίτες να βγουν τα αντίστοιχα συμπεράσματα ε, και να έχει και συνέπειες. Το Συμβούλιο λοιπόν πήρε την απόφαση αυτή που έχει συνέπειες να προχωρήσουμε σε μια τραπεζική ένωση και αυτός ο στόχος βεβαίως αξίζει την υποστήριξή μας και είναι και στα πλαίσια των όσων ήθελε ήδη από τότε το Κοινοβούλιο. Και, εν πάση περιπτώσει, καλή αργά παραποτέ. Τώρα, ε, όμως έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος γιατί η Τραπεζική Ένωση και οι αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνδέονται με το μηχανισμό σταθερότητας. Ε, ε, μετά από αυτές τις ζημιές που πάθαμε όμως θα πρέπει να έχουμε μια δομή που να εποπτεύουμε σωστό τρόπο τις τράπεζες και να λειτουργεί. Και ταυτόχρονα όποιος θέλει να έχει πρόσβαση για χρηματοδότηση ε, από ε, ευρωπαϊκά ταμεία βεβαίως θα πρέπει να ε, υποκλίνεται σε λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι σωστό αυτό, αλλά πώς θα γίνει. Και θα πρέπει να δούμε και το χρονικό πλαίσιο. Δηλαδή επειδή πιέζει ο χρόνος να ε, χρονοτριβεί το Συμβούλιο και εμείς να τρέχουμε. Ήδη το Συμβούλιο έχει βάλει το ίδιο ένα χρονικό πλαίσιο και δηλώνει αδυναμία να ανταποκριθεί σε αυτό. Οπότε εμείς θα πρέπει με την ησυχία μας να τα συζητήσουμε όπως ε, κάνουμε πάντα σε εκθέσεις τα απαραίτητα χρονικά όρια. Λοιπόν, ε, ο εξευρωπαϊσμός, να το πω έτσι, της υποπτίας των τραπεζών έχει πολλούς στόχους. Βεβαίως, αποτελεσματικότητα, ε, όχι επικαλύψεις δομών, ε, σαφήνεια, καλύτερη λειτουργία, δηλαδή πιο ισχυρή ε, ευρωπαϊκή εποπτεία των τραπεζών με ισχυρά δικαιώματα. Ωραία. Αλλά τι σημαίνει αυτό. Ότι χρειαζόμαστε και δημοκρατικό έλεγχο όταν είναι ισχυρά αυτά τα δικαιώματα. Ακόμα και αν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή αν συμπεριλαμβάνεται και η Κεντρική Τράπεζα. Ισχύει ο δημοκρατικός έλεγχος διότι είναι ανεξάρτητη η ΕΚΤ και καλά κάνει. Ε, στην νομισματική πολιτική, αλλά υπάρχει και η δημοσιονομική πολιτική και βασικός δημοκρατικός έλεγχος σημαίνει τα εξή πέντε. Πρώτον, δικαίωμα και με μονομένων βουλευτών να κάνουν ερωτήσεις του δικού μας κοινοβουλίου. Δεύτερον, τακτικές εκθέσεις να λαμβάνουμε και ε, να κάνουμε ερωτήσεις και σε προφορική ανταλλαγή απόψεων. Τρίτον, το δικαίωμα ε, τον εκάστοτε διευθυντή να τον διορίζουμε εμείς Τέταρτο δικαίωμα, να ψηφίζουμε τον προπολογισμό τους. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα και οι ερωτήσεις και οι ακροάσεις θα λαμβάνονται σοβαρά ε, εφόσον εκ των υστέρων πίπτει ράβδος ή έχουμε τουλάχιστον το δικαίωμα. Και να κάνουμε και έκτακτες ε, ε, έρευνες. Τα έχουμε αυτά τα περισσότερα δικαιώματα ε, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουμε εμείς δημιουργήσει, αλλά όχι απέναντι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και αυτό πρέπει να μας απασχολήσει υπάρχουν και περιορισμοί από τη συνθήκη. Με το άρθρο 130 δημιουργείται ένα πεδίο ένταση που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ευρωπαϊκή εποπτεία, δηλαδή να ανεβαίνουμε επίπεδο ε, στην εποπτεία χωρί να συνοδεύεται αυτό από το δημοκρατικό έλεγχο. Επίση, θα πρέπει να υπάρξει ένα διαχωρισμό μεταξύ τη δημοσιονομική και τη νομισματική πολιτική, γιατί αυτά είναι σε σύγκρουση τώρα μεταξύ του. Και τελικά η νομισματική πολιτική δεν θα πρέπει να είναι όμοιρο τη δημοσιονομική και τούμπαλιν. Αυτό ισχύει και για την τραπεζική εποπτεία. Επίσης θα πρέπει να ισχύει εξή αρχή. Μια εσωτερική αγορά θα πρέπει να έχει μια εποπτεία ε, στην οποία να υπόκεινται όλα τα χρηματοπιστωτικά ε, ε, ιδρύματα. <coughs> Αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο. Αν έχουμε μια μικρή τράπεζα τη γειτονιά, ένα ταμιευτήριο στο χωριό, δεν θα πρέπει να έρχονται από τη Φραγκφούρτη, από το Λονδίνο να την ελέγχουν. Αλλά κάποιε μεγάλε τράπεζε που έχουν και πανευρωπαϊκή παρουσία και όταν πάθουν καμιά ζημιά αυτό αφορά όλη την Ευρώπη, ε, θα πρέπει να ελέγχονται κεντρικά. Και όταν κάτι πάει στραβά θα πρέπει το ευρωπαϊκό επίπεδο να έχει τη δυνατότητα παντού όμω να επεμβαίνει. Κάτι άλλο που θα ήταν βέβαια το ιδεώδε. Ένα καθεστώ τέτοιο να συμπεριλαμβάνει όλα τα κράτη-μέλη. Οι εποπτικές μας αρχές το κάνουν αυτό. Αλλά, και έρχομαι τώρα στη δική μου έκθεση, δεν μπορούν να συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη έτσι όπως προτείνεται το σύστημα. Και πολύ χειρότερο όταν υπάρχουν μεγάλες αγορές στις χώρες αυτές που δεν συμμετέχουν. Αυτό δεν είναι αδυναμία αυτή την αδυναμία θα πρέπει να την περιορίσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Γι' αυτό η νέα δομή να γίνει όσο ε, γίνεται πιο ελκυστική για να μπουν όλα τα κράτη-μέλη. Να είναι ένας γλυκός πειρασμός στον οποίο να μην μπορεί κανείς να αντισταθεί παρά με πολύ μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή να μην μπορούν να κάνουν αλλιώς οι χώρες αυτές, να θέλουν οπωσδήποτε να μπουν. Να, μην μπορούν να εξηγήσουν στους πολίτες τους γιατί δεν συμμετέχουν σε αυτό το σύστημα. Και αντίστροφα, θα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ελκυστικό για να έρχονται και άλλε χώρε. Γιατί μπορεί να υπάρξει και ένα διχασμό. Ε, και το να είναι διαιρεμένη η εποπτεία των τραπεζών είναι το χειρότερο που μπορεί κανείς να φανταστεί όταν θέλει μια ε, ουσιαστική οικονομική και νομισματική ένωση γιατί θα δημιουργηθεί προηγούμενο. Και αυτό είναι κακή αρχή για την εσωτερική αγορά. Εμείς ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχουμε ω ρόλο να περιορίσουμε όσο γίνεται περισσότερο αυτό το πρόβλημα. Όλα αυτά που σας λέω, τι σημαίνουν συγκεκριμένα για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα τμήμα των αποφάσεων, ένα τμήμα των αποφάσεων να λαμβάνονται από έκτακτες ειδικέ δομές, ιδιαίτερα ε, για ε, διακανονισμούς διαφορών σε περίοδους κρίσης. Αυτό που θα οδηγούσε. Χρειάζονται διπλές πλειοψηφίες. Και γενικότερα, αλλά και... Πώς να το πω, να το εξηγήσω λίγο. Δημιουργείται μια ξεχωριστή επιτροπή με έκτακτες θέσεις και έδρες που προβλέπονται για αυτούς που δεν συμμετέχουν στη συνεργασία. Και σε περίπτωση που παίρνει αποφάσεις αυτό το πάνελ, στις έκτακτες περιστάσεις και απορριφθούν από το Εποπτικό Συμβούλιο υπάρχει ένα σύστημα διπλής πλειοψηφίας. Δηλαδή, εκτός από τις θετικές ψήφους των χωρών που συμμετέχουν, χρειάζονται και τουλάχιστον τρεις θετικές ψήφοι από τις χώρες που δεν συμμετέχουν. Αυτό βοηθάει τώρα ε, για να λαμβάνονται αποφάσεις, δίνει κίνητρα για ένα μικρό κράτος μέλος να πει ότι Ωραία, θα μπω σε αυτή τη συνεργασία. Και πώς ε, θα την επηρεάζω. Μήπως θα την επηρεάζω περισσότερο απ' έξω. Θα πρέπει να υπάρχει ένα κίνητρο και ε, ένα συμφέρον και για μια μικρή χώρα να μπει σε αυτό το σύστημα παρά να είναι απ' έξω. Το ίδιο ισχύει και με το Διοικητικό Συμβούλιο και πώς ορίζουν τα μέλη του εκεί. Εάν ε, είναι τέτοια η απαρτία θα πρέπει να υπάρχουν πραγματικά τα κίνητρα για να συμμετέχουν οι χώρες. Και έχουν νόημα οι απόλυτοι αριθμοί, ε, ε, αν δεν γνωρίζουμε πόσες χώρες θα μπουν στη συνεργασία. Μπορεί όλες, μπορεί σχεδόν όλες, αλλά οι απόλυτοι αριθμοί είναι πρόβλημα. Αφήστε που αλλάζουν. Κάθε φορά θα πρέπει να τους αλλάζουμε και τους αριθμούς. Δεν γίνεται να βρούμε άλλες λύσεις εκεί. Επίσης, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και ένα δύσκολο ερώτημα, αλλά πολύ ειλικρινά. Μπορεί κανείς να φανταστεί ότι σε περίπτωση διακανονισμού διαφορών σε σημαντικές περιπτώσεις να κάνει προτάσεις η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Δηλαδή αυτή που είναι αρμόδια για το σύνολο της εσωτερικής αγοράς να απευθύνεται σε εκείνη τη μικρή που είναι για ε, τραπεζική ένωση. Είναι περίπλοκο σύστημα. Αυτό θα δημιουργηθεί μεγάλε δυσκολίε. Θα πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό. Λοιπόν, συνοψίζω. Το κοινοβούλιο σε όλο αυτό το θέμα θα πρέπει να είναι ε, υπερασπιστής της συνοχής της Ένωσης των Δημοκρατικών Δικαιωμάτων και θα πρέπει να προσέξουμε. Όχι για λόγους χρονικούς ή για προσχηματικούς νομικούς ας πούμε λόγους να βιαστούμε ε, και να ορίσουμε κάποιους κανόνες που τελικά θα ισχύσουν για την νομισματική ένωση. Έχουμε κάποιες ευθύνες, θα πρέπει να τις ε, αναλάβουμε ε, με την ισχύα μας, με το χρόνο που χρειαζόμαστε και όσο γίνεται με ομοψυχία. Γιατί και στο τελευταίο πακέτο εποπτείας φάνηκε ότι δεν είναι απαραίτητα αυτό που ψηφίζει και αποφασίζει άρον άρον το Συμβούλιο είναι σωστά και ε, ευσταθούν όταν κατεβαίνουν μέχρι τα εθνικά συμφέροντα. Γιατί σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό πνεύμα το Κοινοβούλιο είναι πολύ ισχυρότερο από ότι το Συμβούλιο. Τώρα θα πρέπει να παίξουμε αντίστοιχο ρόλο. Και σε αυτή την περίπτωση χαίρομαι πολύ για τη συνεργασία μου με τη Μαριάν Τάισον και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Γκίγκολτ. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τους σκιώδεις εισηγητές και μετά θα ακούσουμε εναλλακτικά ένα εισηγητή για την έκθεση Tyson και ένα εισηγητή σκιώδη για την έκθεση Γκίγκολτ. Ο κύριος Πιτέλα. Ευχαριστώ πρόεδρε παίρνω το λόγο για την πρόταση κανονισμού σχετικά με το ρόλο της, των κεντρικών τραπεζών, της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας μάλλον. με τις παρατηρήσεις που έκανε ο κύριος Γκίγκολτ. Ήταν πάρα πολύ θετικές και οι εχμές τις οποίες ε, μας παρουσίασε ο κύριος Γκίγκολτ. Είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης η πρότασή του θεωρώ ότι η εποπτεία εφόσον αναλυφθεί από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα είναι κάτι που συνδυάζεται με τις εθνικές αντίστοιχες προσπάθειες και μειώνει ε, τους κινδύνους και σε επίπεδο πιστοτικό και γενικότερα. Υπάρχουν όμως ορισμένα σημεία που πρέπει να συζητηθούν. Το έθεσε εδώ και η κυρία Τίσεν αυτό. Όπως επανειλημμένα έχει υποθεί, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει στο θέμα με βάση το 127 παράγραφος 6 που περιθωριοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα έλεγα η πρόταση αυτή είναι ανεπαρκής. Εμείς καλούμεθα να μην παίξουμε κανένα αποφασιστικό ρόλο. Αυτό είναι ένα σοβαρότατο λάθος και δεν το λέω αυτό ε, γιατί είμαι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για λόγους συντεχνιακούς αλλά θα πρέπει να βασίζεται θα έλεγα κανείς και στην κοινοβουλευτική πείρα που έχει σωρευτεί στο κοινοβούλιο μας τα τελευταία χρόνια στον τομέα αυτό. Δεύτερο σημείο αφορά τις δυσκολίες εναρμόνισης των διαφορετικών παραδόσεων στον τομέα της πιστοτικής εποπτείας στην Ευρώπη. Όπως γνωρίζετε δεν έχουν όλες ε, οι ευρωπαϊκές χώρες δώσει, εμπιστευτεί την εποπτεία στην Κεντρική Τράπεζα. Στην Γερμανία σαν παράδειγμα κεντρικό ρόλο παίζει το Μπαφίν, ένας οργανισμός που εξαρτάται από το Υπουργείο Οικονομικών. Έχουν σημασία αυτές οι διαφοροποιήσεις και δεν πρέπει να υποτιμηθούν. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή στη συζήτησή μας στο άρθρο 5 του κανονισμού που προβλέπει ότι οι εθνικές αρχές οφείλουν να παίξουν κάποιο ρόλο στην προετοιμασία και την εφαρμογή των δράσεων και παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεύτερον, σχετικά με το πόσο ε, τις ευθύνες, την ανεξαρτησία και το υπόλογο σε εισαγωγικά της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας πράγματι είναι υπεύθυνη μπροστά στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επί της ουσίας όμως αυτή η ευθύνη προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πώς θα γίνει πραγματικότητα ε, διαφορετικά με το τι συμβαίνει με το Συμβούλιο το Κοινοβούλιο αποκλείεται από τη διαδικασία διορισμού των αντιπροσώπων και μελών της Επιτροπής Εποπτείας ή του Συμβουλίου Εποπτείας, του Supervisory Board. Εδώ θέλω να τονίσω κάτι. Η πρόταση κανονισμού προβλέπει ότι θα έχει πάρα πολλές αρμοδιότητες και θα μπορεί επίσης να εκχωρεί περαιτέρω αρμοδιότητες ε, με τα δικές του αποφάσεις. Το θέμα λοιπόν του δημοκρατικού ελέγχου στο οποίο στάθηκε και ο συνάδελφος Γκίγκολντ γύρω από τις δραστηριότητες του Εποπτικού Συμβουλίου τίθεται άμεσα και οφείλουμε να εμβαθύνουμε στο θέμα του δημοκρατικού ελέγχου. Thank you. Mr. Balt. Ευχαριστώ κύριος Μπάλτ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει πρώτα να καταλάβουμε τι συζητάμε και τι θα συζητήσουμε τις επόμενες εβδομάδες και μήνες και τι δεν συζητάμε. Ε, είναι προτάσεις για κοινή εποπτεία των τραπεζών. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση. Ίσα ίσα. Εδώ και δύο χρόνια προσπαθούμε ε, να κινήσουμε το Συμβούλιο προς την κατεύθυνση μιας ευρωπαϊκής εγγύησης τραπεζικών καταθέσεων. Και για τα τραπεζικά ιδρύματα, επίσης κάτι αντίστοιχο ζητούμε εδώ και καιρό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για αυτά τα θέματα όμως υπάρχουν ξεχωριστές εκθέσει εκθέσεις και φάκελοι που έχουμε επιτάπητος και θα έχουμε και την ευκαιρία επιπλέον να συζητήσουμε την έκθεση πρωτοβουλίας της Μαριάν Τάισεν για να προβληματιστούμε για το όραμα του μέλλοντος. Βεβαίως και τα δύο θέματα αυτά συνδέονται, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υποκύψουμε στον πειρασμό να ε, αναμειγνύουμε υπερβολικά αυτά τα θέματα. Δηλαδή και στις δύο εποπτικές εκθέσεις να μην ε, δημιουργήσουμε καταστάσεις που δεν έχουν καμία σχέση. Λοιπόν, για την εποπτεία. Καταρχήν πιστεύω η κοινή εποπτεία είναι κάτι πάρα πολύ ευπρόσδεκτο. Η κρίση τα τελευταία χρόνια κατέδειξε σαφέστατα ότι ο πρώτερος ευρωπαϊκός συντονισμός δεν ε, αρκούσε ή δεν άρκεσε για να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στην κρίση. Γι' αυτό δημιουργήσαμε νέες δομές από το 2011. Το ανέφερε ο κύριος ε, Γκίγκολτ και μάλιστα εκτενέστατα. Τώρα, ένας νέος μηχανισμός δεν επιτρέπεται να δημιουργήσει ε, μια επιπλέον εποπτεία, αλλά ενιαία εποπτεία. Ε, δεν θέλουμε ασάφειες ή επικαλύψεις ε, στις αρμοδιότητες. Αυτό θα πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί. Χρειάζεται ένας επιμερισμός εργασίας και καθηκόντων μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής αφενός και του νέου μηχανισμού αφετέρου. Η συμπερίληψη όλων των τραπεζών είναι κάτι επίσης που μας χαροποιεί, αλλά δεν θα πρέπει κανένα από τα μοντέλα, τα τραπεζικά που λειτουργούν σήμερα να ε, βρεθεί σε μειονεκτική θέση. Γι' αυτό θα πρέπει και οι εθνικές εποπτικές αρχές και οι ευρωπαϊκοί να λειτουργούν πάντα και να συνεργάζονται στα πλαίσια της επικουρικότητας το ιδεώδες ποιο θα ήταν. Να ισχύσει ο μηχανισμός αυτός για όλες τις τράπεζες και των 27 κρατών μελών. Αλλά γνωρίζουμε ότι πολιτικά αυτό είναι δύσκολο να επιβληθεί. Οπότε, ειλικρινά προβληματίζομαι και διερωτώμε πόσο αξιόπιστη μπορεί να είναι μια τέτοια υποπτική αρχή που να μην συμπεριλαμβάνει την ένα χρηματαγορά της Ένωσης. που θα ενταχθεί. Ε, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει βεβαίως πραγματογνωμοσύνη, κύρος, φήμη, γνώσεις και ε, στενή διασύνδεση ε, με το Ευρωπαϊκό Σύστημα BSRB. Αλλά θα πρέπει να διατηρηθεί και να διαφυλαχθεί η ανεξαρτησία και από την πολιτική και από την οικονομία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και να μην έχουμε συγκρούσεις συμφερόντων, νομισματικών, ε, χρηματοπιστωτικών και άλλων. Γι' αυτό θα πρέπει να ε, διαχωριστεί το λειτουργικό σκέλος ε, αυτού του μηχανισμού. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή να παίρνει την απόφαση, αλλά για τον έλεγχο να είναι αρμόδια η Κεντρική Τράπεζα. Γι' αυτό χρειάζεται και δημοκρατικός έλεγχος και σε κάθε περίπτωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτό ισχύει και για την κατεύθυνση που θα πάρει, για τη δημιουργία του μηχανισμού εποπτείας και για τη λειτουργία του. Για μένα είναι αυτό ένα βήμα ενοποίησης αλλά χρειάζεται τη σύμφωνη γνώμη ενός δημοκρατικά εκλεγμένου και νομιμοποιημένου ε, οργάνου. Ε, επανειλημμένα έχουμε τονίσει και πιστεύω προσωπικά θα συνεχίσουμε να το κάνουμε ότι απόφαση για τον πυρήνα ε, της νέας δομής σε επίπεδο συμβουλίου δεν αρκεί. Από την αρχή αμφισβητήθηκε ε, η νομιμότητα της Ευρωπαϊκής ε, Τραπεζικής Ένωσης. Έτσι κι αλλιώς ο πολίτης ε, ήδη αφισβητεί το ίδιο το νόημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε δεν έχει νόημα να πιεζόμαστε από χρονικού περιορισμούς. Δεν είναι μια γρήγορη λύση τώρα για την κρίση των κρατών που αντιμετωπίζουν προβλήματα χρέους. Βεβαίως, ε, είναι το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, αλλά χρειάζεται και ε, ε, μια εποπτεία που να λειτουργεί, όχι που να έχει αποφασιστεί απλώς. Δεν αρκεί μέχρι το τέλος του έτους να ολοκληρώσουμε την νομοθετική διαδικασία, κάτι που είναι πολύ φιλόδοξο από μόνο του, αλλά πρέπει να δημιουργηθούν οι απαραίτητες δομές. Οι πρώτες τράπεζες από την 1η 1 του 2013 ε, για να μπουν στο σύστημα μου φαίνεται πάρα πολύ ε, ανεδαφικό. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα και από το ΕΚΟΦΗΝ που ε, ε, αφιερώθηκε σε αυτό το θέμα. Σταματώ εδώ, θα είχα πάρα πολλά να πω ακόμα, αλλά για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και μια πρώτη επισκόπηση αρκεί. Ευχαριστώ πολύ. Mr. Ευχαριστώ κύριος Κλίντς. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Όλοι οι προλαλήσαντε ξεκαθάρισαν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όχι απλώς καλωσορίζει αυτό, αυτή την πρόταση, αλλά τη ζητούσαμε εδώ και δύο χρόνια. Και μάλιστα πολύ πιο ισχυρή αποπτία από αυτή που μας προέκυψε ε, τελικά. Το ερώτημα όμω τώρα που τίθεται είναι, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να ενταχθεί αυτή η δομή. Διότι τότε εμείς λέγαμε να είναι κάπου κοντά στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά όχι απαραίτητο υπό τη στέγη της ΕΚΤ. Να υπάρχει ένας διάλογος, πολύ σημαντικός βεβαίως με την εποπτική αρχή, αλλά εάν την εντάξουμε στις δομές της Κεντρικής Τράπεζας υπάρχουν εξή δύο κίνδυνοι. Πρώτη, κάποια στιγμή θα πάει κάτι στραβά και οι επόπτες κάνουν λάθη και εκεί διακινδυνεύουμε την αξιοπιστία, ε, το κύρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επίσης είπαμε ότι η θέλουμε να είναι ανεξάρτητη και να εξακολουθεί να είναι αρμόδια για την νομισματική πολιτική. Και θα υπάρξει η περίπτωση, ε, σε περίπτωση κρίσης, να χρειαστούν χρήματα για να σωθούν ή να στηριχτούν τράπεζες ε, σε εποχή που ο μηχανισμός σταθερότητας δεν είναι ακόμα ε, στα πόδια του ούτε λειτουργεί, ε, διότι θα χρειαστούν και χρόνια για να γίνει αυτό. Οπότε ε, είναι θέμα των χρημάτων των φορολογουμένων, βλέπε Υπουργοί Οικονομικών, βλέπε πολιτική. Λοιπόν, μια τέτοια αρχή εποπτική το να δρά υπό πολιτικές πιέσεις Υπουργών Οικονομικών δεν μπορεί να είναι κάτι που εμείς επιθυμούμε. Και όταν συζητούμε για εποπτεία, θυμάστε τι είχαμε πριν από δύο χρόνια αρκεί να δημιουργήσουμε μόνο για τις τράπεζες Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή. Γιατί οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι πολύ κοντά. Κάτι λέει ο κύριος Λάγκεν εκτός μικροφώνου. Α, τη συνθήκη, τη συνθήκη. Ναι, το ξέρω ότι είναι η συνθήκη Βέρνερ. Γι' αυτό ε, ρωτώ αν θα πρέπει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να γίνει δίπλα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να είναι αρμόδια αυτή η αρχή όχι μόνο για τις τράπεζες αλλά και για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Για το μέλλον μου φαίνεται αυτό καλύτερο. Οι προλύσαντες αναφέρθηκαν σε πολλά ζητήματα και με τις τοποθετήσεις τους συμφωνώ, όχι μόνο συμφωνώ, τις καλωσορίζω και τις χαιρετίζω σε μεγάλο βαθμό και βέβαια έχουμε συμφέρον ε, να μην διχαστούμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατανοώ ότι υπάρχουν καθεστώτα που χρειαζόμαστε και συστήματα για την Ευρωζώνη για να σταθεροποιήσουμε το νόμισμά μας. Εντάξει, αλλά δεν θα πρέπει να διαιρέσουμε τώρα έτσι την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε και το λέω άμεσα οι Βρετανοί να ενθαρρυνθούν και να πούνε σε ένα δημοψήφισμα ε, παιδιά φτάνει και βγαίνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. That's it, τελειώσαμε. Ε, αυτό οπωσδήποτε θα πρέπει να το αποφύγουμε και να το αποτρέψουμε. Λοιπόν, πώς θα γίνει αυτό. Οι πρακτικοί ε, μηχανισμοί λήψης αποφάσεων πρέπει να είναι έτσι ορισμένοι και με τις αρμοδιότητες που να λειτουργούν σωστά. Υπόθηκαν από τους προλήσαντες, θα πρέπει, προσοχή, ε, να μην δημιουργήσουμε δομές λήψης αποφάσεων που τελικά μάλλον δρούν ως αντικίνητρο εγώ θα πρότεινα το εξή. Όλα τα κράτη που αποφάσισαν να μπουν στην Ευρωζώνη, που έχουν ζητήσει και 25 με εξαίρεση τη Μεγάλη Βρετανία και τη Δανία, ε, θα πρέπει να μπουν σε αυτό το σύστημα, γιατί είναι και νομικά δεσμευτικά αυτά με βάση και το διεθνές δίκαιο, έτσι δεν είναι. Ζητήσατε κάποια στιγμή να μπείτε, δεν ξέρω, ίσως και στο απότερο μέλλον, ε, να μπείτε στην ΟΝΕ, ναι, οπότε μπορείτε να μπείτε και στο σύστημα από τώρα. Παρ' όλα αυτά το μέγα πρόβλημα παραμένει ότι η μεγαλύτερη χρήματα αγορά ε, και ε, χρηματοπιστωτική έδρα το Λονδίνο μένει εκτός. Ε, αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε για να μην κάνουμε καμιά ζημιά. Άλλο θέμα τώρα. Βεβαίω η αρχή τη επικορικότητα και της αναλογικότητα πρέπει να γίνουν σεβαστέ. Θα πρέπει να έχει την αρμοδιότητα αυτή η δομή να ελέγχει όλες τις τράπεζες της Ευρωζώνης ή των χωρών που συμμετέχουν. Αυτά είναι στη θεωρία. Στην πράξη όμως θα γίνει αυτό ε, μέσω της αντιπροσωπείας της Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές. Παράδειγμα, μικρά ταμιευτήρια, μικρέ ιδιωτικέ τράπεζε υπάρχουν στη Γερμανία. Δεν μπορούν να ελέγχονται έτσι στην καθημερινή του λειτουργία, να επιθεωρούνται από αυτή τη μεγάλη δομή. Υπάρχει μια τράπεζα που λέγεται Castell Bank, είναι σαν μεγάλο τραμευτήριο και δρεύει στο Würzburg ε, και είναι ιδιωτική τράπεζα. Εάν τεθεί το ζήτημα τη αφαιρηθεί λειτουργίας, ποιο θα το λύσει αυτό, η Ευρωπαϊκή Αρχή. Ναι, αλλά ε, στην ε, καθημερινή δραστηριότητα θα ελέγχει η αρμόδια γερμανική αρχή που λέγεται Μπάφιν. Λοιπόν, ενιαία εποπτεία, αναδιάρθρωση και καθάριση και ένα σύστημα εγγύησης των καταθέσεων. Τώρα, το ταμείο αυτό που θα πρέπει να λειτουργεί σε διάφορα κράτη-μέλη για την αναδιάρθρωση και για τις εκαθαρίσεις θα πρέπει ε, να ε, λειτουργεί ενιαία, όχι όπως γίνεται σήμερα. ότι ε, το θέμα της εξαγοράς τραπεζών ή της μεταβίβασης σε κάθε χώρα δεν ρυθμίζεται με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες, διαφορετικές καταστάσεις. Ε, για να τα λύσουμε όλα αυτά, για να δημιουργηθεί ένα ενιαίο ταμείο, θα χρειαστεί μια δεκαετία για να έχει και ένα ποσό σοβαρό και να μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση σε περίοδους κρίσης. Λοιπόν, έχουμε συζητήσει με τους σκιώδεις συζητητές, παραμένουμε στην πρότασή μας, να παραμείνει αυτό στα χέρια των εθνικών ε, ρυθμιστικών αρχών. Έχω ακόμα πολλά θέματα, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί τα είπαν οι προηγούμενοι μιλητές, αλλά ένα τελευταίο. Η δημοκρατική νομιμοποίηση και η ε, λογοδοσία. Τώρα πώς έχει η κατάσταση η δομή αυτή και η θεσμική δομή και η διαδικασία λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται όλο και πιο περίπλοκη και πιο θολή. Ο πολίτη δεν καταλαβαίνει πια πώ λειτουργεί η Ευρώπη. Και αυτά που κάνουμε τώρα με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική από τη μια αρχή και από την άλλη την εποπτεία στην Κεντρική Τράπεζα δεν βοηθάει τον κόσμο, δεν διευκολύνει τα πράγματα. Γι' αυτό έχουμε το καθήκον και την υποχρέωση να εξασφαλίσουμε ότι ο πολίτης να μπορεί να απευθύνεται τουλάχιστον σε εμά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να βλέπει σε εμά ένα όργανο το οποίο ανταποκρίνεται στο χρέος του και ελέγχει δημοκρατικά τις νέες δομές. Και ισχύει και αυτό που είπε και ο Γκίγκολτ. Τώρα, ε, από εκεί και πέρα ένα κοινοβούλιο έχει πάντα το ρόλο να εκπροσωπεί τον κυρίαρχο λαό. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Σας ευχαριστώ κύριε Κλίντς. Ο κύριος Πρεσέντο συμφώνησε ήδη να πάρει το λόγο μετά από τον κύριο Λάμπερτ που πρέπει να φύγει. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ επίσης τον, τον Ιν που με αφήνει να πάρω το λόγο νωρίτερα. Στα γαλλικά λέμε ότι δεν πρέπει πρέπει κανείς να βιάζεται για σκοντάφτει σκοντάφτη ε, και βιαζόμενοι να φτάσουμε σε πορίσματα μπορεί να φτιάξουμε ένα οικοδόμημα το οποίο να είναι σαθρό. Και άκουσα διάφορο στο Συμβούλιο να λένε ότι πρέπει να το καταφέρουμε αυτό σωστά. Και συμφωνώ με αυτό και το γεγονός ότι έχουμε καταστήσει αυτό προϋπόθεση για την άμεση ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών είναι κάπως ατυχές διότι δημιουργούμε λάθος κίνητρα νομίζω για το να δράσουμε τελικά με σωστό ή λάθασμένο τρόπο. Θέλω να επανέλθω στα όσα είπε εσύ, Μαριάν, ότι δηλαδή αναγνώρισε τη δήλωση του Συμβουλίου που επανελήφθη πρόσφατα ότι πρέπει δηλαδή όλα αυτά να το αναθέσουμε στην έκτο, ότι αυτό μπορεί να έχει πλέον χτήματα αλλά και περιορισμού. Και με βάση τα όσα είπε ο Σβέν, θέλω να πω τα εξή. Πρώτον, ισχυρή δημοκρατική λογοδοσία. Δεύτερον, ίση συμμετοχή για τα μέλη και τα μη μέλη του ευρώ. Δεν θέλουμε να έχουμε δηλαδή δύο διαφορετικές τάξεις συμμετεχόντων. Το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι κατά πόσο οι ισχύοντες νομικοί περιορισμοί που συνδέονται με την ΕΚΤ μας επιτρέπουν να κάνουμε σωστή δουλειά για αυτά τα δύο πράγματα. Δηλαδή, είτε θα πούμε είναι η ΕΚΤ, δεχόμαστε τους περιορισμούς και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε όσον αφορά την ίση συμμετοχή και τη δημοκρατία μέσα σε αυτά τα όρια, ή θα πούμε όχι. Το όριο είναι η δημοκρατική λογοδεσία και η ίση συμμετοχή. Αυτές είναι οι αρχικοί όροι και έπειτα κατά πόσο, με βάση το κατά πόσο η ΕΚΤΕ θα μπορέσει να μας δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα, θα πάμε εκεί ή θα αναζητήσουμε εναλλακτικέ. Εγώ πιστεύω πως χρειαζόμαστε πολύ στεναρή νομική συμβουλή στις αρχές. Όχι στο τέλος, όταν θα έχουμε ένα πολύ ωραίο οικοδόμημα και έρθουν νομικοί και μας πούνε «Μπράβο παιδιά», αλλά αυτό δεν πρόκειται να λειτουργήσει μέσα στους περιορισμούς αυτούς, γιατί μετά θα ασκηθεί πίεση για να πούμε ότι παρόλα αυτά θα το προχωρήσουμε και να έχουμε δηλαδή έτσι χειρότερες λύσεις, δηλαδή κάτω από τα, τις προδιαγραφές. Να πω κάτι ακόμα. Το Κοινοβούλιο μας ζητά ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή εποπτεία όχι μόνο των τραπεζών αλλά και των ασφαλιστικών και των ε, χρηματοπιστωτικών αγορών και ξέρουμε πως όλα αυτά τα τρία είναι πολύ πολύ στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι λοιπόν στις τράπεζες ε, στο ΕΝΕΚΤ που θα μας εμποδίσουν από το να, ολοκληρώσουμε, να, να επιτύχουμε την ολοκλήρωση που θέλουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ας πούμε, απαγορεύεται ο ρόλος, ε, άσκηση μάλλον ρόλου της ΕΚΤ στις ασφαλιστικές. Τι κάνουμε λοιπόν με τους ομίλους, τους αφήνουμε ήσυχους Θέλουμε να, να φτιάξουμε, όχι να κάνουμε μια ανακαίνιση ενός κτίριου, αλλά να κάνουμε μια επέκταση του ίδιου κτίριου. Και επειδή ξέρουμε εξ αρχής ότι δεν θα μπορέσουν να υπάρξουν επεκτάσεις προς την ε, κατεύθυνση των ασφαλιστικών ή των χρηματοπιστωτικών αγορών, αυτό θα πρέπει από την αρχή να το συνειδητοποιήσουμε και να μην πούμε αργότερα «Ωχ, παιδιά, εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα» προς αυτές τις κατευθύνσεις. Λοιπόν, δεν θέλω να βιαστώ να φτάσω σε συμπεράσματα, αλλά πρέπει εξ αρχής να καταλάβουμε ποιοι είναι οι περιορισμοί της επιλογής που θα κάνουμε. Ε, γιατί πιστεύω ότι στο Συμβούλιο ορισμένοι αρχίζουν να το ξανασκέφτονται. Και άρα δεν είναι θέμα του να κρατήσουμε το γόητρό μας, αλλά καταλάβουμε ότι λάθος προχωράμε, θα πρέπει ε, να, ενεργήσουμε διαφορετικά. Αλλά δεν... νομίζω ότι θα πρέπει να δουλέψουμε μόνο πάνω στα όρια τα οποία έχει θέσει το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ. Τώρα ο κύριος Πρεζέντο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους και ε, και τους δύο παρόλο που είναι δύο διαφορετικές πρωτοβουλίες, είναι πακέτο η πρόταση αυτή. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένα τα δύο μεταξύ του. Οπότε, η πρόταση για την κεντρική τράπεζα ε, θα μπορούσε το ένα να είναι μια πρόταση κανονισμού για την αλλαγή ε, της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής και το άλλο στην απόφαση. Αλλά ε, θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να έχουν τη βεβαιότητα ότι ε, θα ληφθεί απόφαση με βρία συνένεση και ομοφωνία. Είναι λοιπόν ενιαίο το πακέτο. Όταν συζητούμε την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Εποπτεία και στο παρελθόν ξέραμε όλοι ότι έχει περιορισμούς η πρόταση. Τότε λέγαμε όταν δεν υπάρχει ένα σύστημα αγγίσης καταθέσεων, ένα μηχανισμός ε, καθάρισης ευρωπαϊκός, δεν βοηθούσε. Και θα βοηθούσε αν δημιουργηθεί αυτό για μια ευρωπαϊκή εποπτεία. Περάσαμε λοιπόν από μια ε, συνεργασία ε, μια συνεργασία και νομοθεσία από της αρχής, αλλά αφήναμε στην άκρη τα πρακτικά ζητήματα. Τώρα έχουμε προχωρήσει περισσότερο στα τεχνικά, στην εφαρμογή. Θεσπίσαμε μηχανισμούς για να λύνουν ε, διαφορές σε έκτακτες καταστάσεις και ένα σύστημα ευρωπαϊκής εποπτείας. Είναι όμως προφανές και αυτονόητο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προχωρήσει ακόμα περισσότερο Δηλαδή είναι υπαρξιακό το, ζήτημα, για την Ευρωζώνη. Επίσης δεν θα πρέπει να αποκλείεται κανένας άλλος για να μπορούν να συμμετέχουν και τα άλλα κράτη-μέλη. Η Ευρωζώνη δημιουργήθηκε μετά από συμφωνία δημοσιονομική, αλλά χρειάζεται και χρηματοπιστωτική. Γιατί τελικά τα ε, δημόσιο-οικονομικά, τα χρηματοπιστωτικά είναι αυτά που συνδέουν την νομισματική πολιτική με την πραγματική οικονομία. Πρέπει δηλαδή να προχωρήσουμε πιο πέρα. Εχθές ε, σε μια ομιλία του στο Βερολίνο ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είπε ότι ο μηχανισμός που διαθέτει η τράπεζα για να εξασφαλίζει τη σταθερότητα των τιμών είναι το κόστος του ε, δανείου. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει ενιαίο νόμισμα ε, και αναοικογένεια ή αναεπιχείρηση να έχεις διαφορετικό κόστος για δανειοδότηση και δεν μιλώ για κράτη εδώ. Γι' αυτό χρειάζεται ε, τραπεζική ένωση η Ευρωζώνη για υπαρξιακούς καθαρά λόγους και για το <coughs> κόστος των δανείων για να μην έχουμε αυτές τις ε, κούρσες και τη διαρροή κεφαλαίων από τη μια χώρα στην άλλη και για να λυθεί επίσης ε, με λογικό τρόπο αυτό το θέμα επιλύσει της κρίσης χωρίς να υπάρχει ηθικός κίνδυνο και χωρίς να την πληρώνουν τελικά οι ε, πολίτες. Και ε, ε, τώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προτείνεται με ΑΙ ως αρχή στην οποία θα ενταχθεί η Τραπεζική Ένωση. Νομίζω ότι είναι λογική η πρόταση αυτή, διότι στα περισσότερα κράτη-μέλη ε, συμφωνούν με αυτή την πρόταση και εμείς οι ίδιοι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουμε δώσει ένα ρόλο μακροεποπτείας. Δηλαδή ήδη έχουμε δημιουργήσει προηγούμενο για το πώς θα συνδέονται οι διάφορες αρμοδιότητες υποπτίας. Υπάρχουν εδώ διαφορετικά και διάφορα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Το ένα είναι ο επιμερισμός και ο διαχωρισμός των καθηκόντων. Δεν είναι το ίδιο η προληπτική εποπτεία με την νομισματική πολιτική. Η προληπτική εποπτεία έχει ε, να κάνει ε, και με τη δανειοδότηση νοικοκυριών, οικογενειών και επιχειρήσεων Υπάρχουν διαφορετικοί μηχανισμοί για κάθε ε, κατάσταση, άλλο Ευρωζώνη, άλλο οι χώρες εκτός Ευρωζώνης. Ο διαχωρισμός λοιπόν των λειτουργιών θα πρέπει να είναι σαφής και επιπλέον σε ό,τι αφορά την εποπτεία θα πρέπει να υπάρχει πλήρης δημοκρατικός έλεγχος από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τον ίδιο τρόπο που ισχύει σε οποιοδήποτε από τα κράτη-μέλη μας. Εδώ νομίζω συμφωνούμε. Για την περίμετρο της Τραπεζικής Ένωσης. Δύο στοιχεία. Σε ποιες τράπεζες θα αναφέρετε. Εγώ νομίζω όλες. Σε όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Γιατί είδαμε ότι οι συστημικοί κίνδυνοι δεν έρχονται μόνο από τι μεγάλες τράπεζες. Πολλές φορές είναι η ανάληψη πολλών κινδύνων από μικρές ε, τράπεζες. Και ταυτόχρονα ε, θα πρέπει να έχουμε κανόνες παιχνιδιού ε, ίδιους για όλους. Επίσης, με τον ίδιο τρόπο ε, θα γίνεται και όλες οι εθνικές αρχές θα συμμετέχουν αλλά δεν θα λειτουργούν ως εθνικές αρχές, αλλά ως ένα τμήμα μιας ευρωπαϊκής δομής εποπτικής. Και βεβαίω οι πρακτικέ μπορεί να συνεχίσουν ακριβώ οι ίδιε, αλλά αυτό που θα αλλάξει θα είναι η δομή και ο τρόπο οργάνωση και ε, τη εποπτεία και η διάστασή τη. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι πώ συνδέεται η Τραπεζική Ένωση με τι χώρε που δεν είναι μέλη του ευρώ. Εκεί πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε τρόπους για να συμμετέχει το Κοινοβούλιο. Η Τραπεζική Ένωση είναι εκ των όνων άνευ αλλά χρειάζεται και μια συνεργασία με τα κράτη-μέλη που θέλουν να συμμετέχουν. Αυτό ενισχύει την εσωτερική αγορά και ε, θα πρέπει να βρούμε κάποιο μηχανισμό να διαρθρωθεί έτσι το σύστημα ώστε να μπορούν και χώρες εκτός Ευρωζώνης να συμμετέχουν. Επίσης πρέπει να πω και θέλω να πω ότι συμφωνώ με όλα όσα υπόθηκαν για την ανάγκη εντατικοποίησης της ε, δημοκρατικής νομιμότητας, ε, της εποπτείας και της Τραπεζικής Ένωσης και να ε, διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο το Κοινοβούλιο εκεί. Από τώρα, από το πακέτο αυτό και τη συζήτηση που πρέπει να ειδωθεί ως ενία δέσμη πρόταση και από την αρχή να αντιμετωπιστεί ως ενία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η κυρία Γκουλάχ. Α, έφυγε η κυρία Γκουλάχ. Ο κύριος Τρίτσεκ, σκιώδης για την πολιτική του ομάδα και στις δύο αυτές εκθέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Eh, já myslím, Η συζήτηση που γίνεται τώρα είναι πάρα πολύ χρήσιμη και είναι σωστό το ότι αντιμετωπίζουμε και τις δύο εκθέσεις από κοινού. Οι ιδέες που ακούστηκαν γύρω από τις εκθέσεις Γίγκολντ και Τάισεν... Ε, θα έλεγα δείχνουν ότι τα θέματα αυτά είναι φυσικά παράλληλα. Διαπιστώνω εδώ ε, γύρω μου ότι όλες οι πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, αντιμετωπίζουν το ίδιο δίλημα με τους Ευρωπαίους συντηρητικούς. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από χώρες στην Ευρωζώνη και από χώρες οι οποίες είναι εκτός Ευρωζώνης. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίζετε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και εμείς. Εγώ σαν σκιώδης ε, εισηγητής ε, θα πρέπει να αντιπροσωπεύω τον κύριο Έπινγκ σαν παράδειγμα, τον συνάδελφο Έπινγκ ο οποίος είναι ε, μέλος η χώρα του της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί του ότι για τη δική του χώρα η εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι η καταλληλότερη λύση για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Όμως αυτό ισχύει για αυτόν και αυτό ισχύει και για τους άλλους εκπροσώπους χωρών μελών της Ευρωζώνης. Το θέμα βέβαια και για αυτούς είναι το πόσο ισχυρή θα είναι αυτή η εποπτική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η συζήτηση λοιπόν γύρω από τον ενιαίο ευρωπαϊκό μηχανισμό είναι μια συζήτηση η οποία θεωρητικά είναι εύκολη. Το θέμα είναι όμως η εμβέλειά της αυτής της αρχής. Θα καλύπτει το σύνολο της Ευρωζώνης, ε, θα καλύπτει την Ευρωζώνη και αυτούς που έχουν ζητήσει να μπουν στην Ευρωζώνη θα είναι υπεύθυνη η εποπτική αυτή αρχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς αυτές είναι συζητήσεις που δεν έχουν ε, ολοκληρωθεί. Εμείς που είμαστε εκτός των 17, εκτός Ευρωζώνης, θεωρούμε ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές θα πρέπει να διατηρήσουν πλήρως τις αρμοδιότητές τους. Και τίθεται εδώ το θέμα και τι αρμοδιότητες θα απομείνουν στις εθνικές εποπτικές αρχές. Ποιος θα έχει την τελευταία λέξη. Ένα πράγμα είναι να αναφέρεται κανείς στις εξουσίες της κεντρικής αρχής και ένα άλλο θέμα είναι να σεβαστεί κανείς τις συνταγματικές ρυθμίσεις της κάθε χώρας έχουν κάποια όρια και κάποιους ρόλους να παίξουν οι εθνικές εποπτικές αρχές ανάλογα με αυτά τα οποία προβλέπει το Σύνταγμά τους. Και είναι υπόλογες αυτές οι εποπτικές αρχές σύμφωνα με το Σύνταγμά τους για την οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα της χώρας τους. Αυτό δεν είναι δεν είναι πραγματικά κάτι το οποίο μπορούμε να ξεχάσουμε. Εγώ δεν συμφωνώ πολύ συχνά με τον κύριο Λαμπέρτα αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά έχει δίκιο. Εδώ τίθεται ένα σοβαρό θέμα. Και νομίζω ότι ναι, μεν πρέπει να πάμε γρήγορα, αλλά η βιασύνη είναι κακό σύμβουλος και απαιτείται περισσότερος χρόνος στην επεξεργασία του θέματος. Έχω και κάποια επιπλέον θα έλεγα ελάσσονα θέματα σαν παράδειγμα για τον κύριο Γκίγκολντ. Ο κύριος Γκίγκολντ αναφέρθηκε στην στο πόσο δημοκρατικά θεμητό και πόσο νομιμοποιούμενο δημοκρατικά είναι ε, η διαδικασία την οποία ακολουθούμε και αναφέρθηκε αν κατάλαβα καλά αυτά που είπε σε πέντε βήματα. Εγώ δεν θα ήθελα να πω αν έχει δίκιο ή αν κάνει λάθος ο κύριος Γκίγκολτ. Έχουμε όμως εδώ τη βάση για περαιτέρω συζητήσεις και αναλύσεις. Το δέχομαι αυτό. Ένα δεύτερο επιμέρους και αυτό θέμα ο υπερεθνικός αυτός εποπτικός μηχανισμός θα απαιτήσει αλλαγές στις συνθήκες και μπορούμε να αλλάξουμε τις συνθήκες μόνο εάν τα κοινοβούλια των κρατών μελών είναι σωστά ενημερωμένα. Κανένα δεν αναφέρθηκε στη συζήτηση που έγινε μέχρι σήμερα εδώ, σήμερα το πρωί, στα κοινοβούλια των κρατών μελών. Οι πολίτες των κρατών μελών θα πρέπει να μπορούν να αποφασίσουν μέσω των κοινοβουλίων τους. Αυτό είναι κομβικό. Εγώ δεν λέω ναι ή όχι στην Τραπεζική Ένωση, θα πρέπει οι χώρες, οι πολίτες, τα κοινοβούλια να το αποφασίσουν. Mm, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το δικαίωμα ψήφου μέσα στην Ευρωπαϊκή Εποπτική ε, Τραπεζική Αρχή θα είναι ισορροπημένο ανάμεσα σε, δηλαδή σε αυτούς που είναι εντός του μηχανισμού και εκείνους που δεν είναι. Η εκτός μηχανισμού θα είναι το πιο αδύναμο σκέλος και άρα αν θα πρέπει να φεύγουν κάθε φορά και να μην συμμετέχουν στην ψηφοφορία, όπως και ορισμένοι από σας ήδη είπατε, θα υποβάθμιζε αυτό την ε, διαδικασία ολοκλήρωσης και κάτι τέτοιο θα ήταν απαράδεκτο και δεν νομίζουμε πως θα πρέπει να γίνει, να υλοποιηθεί. Η κυρία Τάισαν νομίζω πως γνωρίζει τους κινδύνους που σχετίζονται με την ε, ανάθεση περισσότερων εξουσιών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διότι ανέφερε και τη σημασία των εθνικών εποπτικών αρχών. Και ακριβώς αυτό είναι το θέμα κλειδί. Ότι δηλαδή ε, όσοι προερχόμαστε από χώρες όπου δεν υπάρχει το ευρώ και έχουμε εθνικές εποπτικές αρχές, θα χρησιμοποιήσουμε τις τροπολογίες ώστε να εξασφαλίσουμε πως στις χώρες μας η εθνική εποπτική αρχή θα έχει τον τελευταίο λόγο. Και αν μου επιτρέπετε να κάνω και ένα τελευταίο σχόλιο, Προτείνω ότι στην συζήτηση για τον ενιαίο επιπτικό μηχανισμό να μην εστιάσουμε σε αυτό ως ένα μεμονωμένο φαινόμενο, θα πρέπει να συνοδεύεται από την Νομισματική και Οικονομική Ένωση, η οποία δεν νοείται ανευπολιτικής ένωσης. Πολιτικές λοιπόν αρμοδιότητες του κέντρου θα πρέπει να ενισχυθούν και αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε εν γέννη γιατί θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω συνοδευτικά μέτρα που θα οδηγήσουν σε στενότερη Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό και ε, επιμένουμε για μια δημοκρατική εντολή που θα συνοδεύει αυτή τη διαδικασία. Ο κόσμος, στα κράτη-μέλη, οι λαοί είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να αποφασίσουν την κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθεί η ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Λήψης Αποφάσεων. Αυτή είναι η απόψη μου και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κλούτε που είναι επίσης εισηγητής, σκιώδης εισηγητής για τις δύο εκθέσεις. Ευχαριστώ. Έχουν υποθεί πολλά. Ε, δεν θέλω να μακρηγορήσω. Γενικά συμφωνούμε δεν έχω να πω τίποτα που να πηγαίνει σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Πρώτον, την Τραπεζική Ένωση το θεωρώ και σκόπιμη και ε, χρήσιμη γιατί δεν μπορεί να έχει κανείς ε, μια αγορά χωρίς τελικά να υπάρχει κοινή εποπτεία και ρύθμιση των τραπεζών. Αλλιώς πάνε στραβά κάποια πράγματα, το έδειξε και η κρίση. Το θέμα είναι όμως πώς θα το διοργανώσουμε όλο αυτό το σύστημα. Και αναφέρθηκαν τα σημαντικότερα σημεία. Προσωπικά έχω κάποιες επιφυλάξεις η εποπτεία να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ακούστηκαν οι λόγοι. Στην έκθεση Giggold φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα ήδη από τη διατύπωση ε, για το πώς θα υπάρξει εκεί το παιχνίδι και ε, η δομή ΕΜΠΑ και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν είναι μόνο οι δομέ, είναι και θέμα προσωπικότητων ε, που πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ του και να μπορούν να συνεργάζονται. Και μπορεί κανεί να φανταστεί τι προβλήματα, τι προστριβέ μπορεί να δημιουργηθούν και ότι είναι πάρα πολύ εκρηκτική η διάρθρωση έτσι όπως την προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπάρχει κίνδυνος αποτυχίας. Για μένα είναι μεγάλο το ερώτημα αυτό, εάν έχει τόσο πολύ νόημα ε, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εντάξουμε και άλλη εποπτική αρχή, πέρα από τις άλλες τρεις που έχουμε. Γιατί αυτό πολλαπλασιάζει τα προβλήματα και συντονισμού και στα διάφορα επίπεδα συντονισμού με τα κράτη-μέλη, έτσι δεν είναι. Αυτό παραμένει ανοιχτό και αναπάντητο ερώτημα. Ε, νέα ρύθμιση για τη ε, όλη λειτουργία βεβαίως και να συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλλά πώς θα γίνει αυτό, Ευρωζώνη και μη Ευρωζώνη. Έχουμε μια νέα αγορά εσωτερική. Είναι συστηματικό το πρόβλημα. Στην έκθεση πρωτοβουλία της Μαριάν Τάισεν ε, γράφει κάτι που συμφωνώ ότι θα πρέπει να αποφεύγεται το αρμπιτράζ στην ε, ρύθμιση αλλά ε, και οι επικαλύψεις και οι συγκρούσεις. Τώρα ανοίγουμε τις θύρες με την πρόταση αυτή, όμως δεν είναι τόσο εύκολο να την αποφύγουμε. Αυτή την κατάσταση γι' αυτό διατηρώ τις επιφυλάξεις μου να μπει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα κάνω και κάποιες τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή, όχι στην ΕΚΤ αλλά στην ΕΜΠΑ, την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Κάτι άλλο ε, το οποίο συμφωνώ είναι αυτό που είπε ο κύριος Μπάλτ. να μπουν όλες οι τράπεζες. Βεβαίω με κάποια κλιμάκωση, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί όλα τα μοντέλα τραπεζών που έχουμε Έχουμε συνεταιριστικές τράπεζες, ταμιευτήρια, μικρές ιδιωτικέ τράπεζε, πολύ σταθερές που άντεξαν στην κρίση. Δεν θα πρέπει να ε, μπουν στο ίδιο τσουβάλι ε, με τράπεζες που εμφάνισαν κάποιες αδυναμίες ε, στην κρίση. Δεν θα πρέπει να καταστρέψουμε κάποιες καλές δομές που λειτουργούν. Δημοκρατικός έλεγχος, λογοδοσία στο κοινοβούλιο, σαφέστατο δεν μπορώ παρά να το υπογραμμίσω, δεν χρειάζεται να επεκταθώ. Ένα μεγάλο ερωτηματικό επίσης για μένα είναι το εξής. Ε, όλη ε, αυτή η ιστορία του παράλληλου τραπεζικού συστήματος, shadow banking, Δηλαδή τι νόημα έχει να ρυθμίζουμε πάρα πολύ καλά και να κλειδώνουμε τις τράπεζες, αλλά υπάρχουν πάρα τράπεζες. Ε, μια παραοικονομία, ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα παράλληλο που να εκφεύγει όλο αυτού του συστήματος ε, και να υπονομεύει τα, ε, όλα καλά και ωραία που έχουμε οικοδομήσει. Αυτά. Τα πρώτα μου σχόλια και σταματώ εδώ. Thank uh, Σας ευχαριστώ. Έχουμε τώρα ένα κατάλογο οκτώ συναδέλφων που ζήτησαν το λόγο. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αλλά και γι' αυτό θα σας παρακαλέσω να είστε σύντομοι. Επίσης η κυρία Γουλάρη είναι σκιώδης. Α, ήρθατε. Ωραία λοιπόν, πάρτε αμέσως τώρα εσείς το λόγο αν είστε έτοιμοι, εκτός αν θέλετε να πάρετε μια ανάσα και να πάρετε το λόγο στο τέλος. Όχι, δεν θέλω να σας ε, ενοχλήσω, είναι λάθος μου, ε, έπρεπε να απαντήσω σε ένα τηλεφώνημα. Θέλω να μιλήσουν οι συνάδελφοι, εγώ θα πάρω το λόγο στο τέλος. Μάλιστα. Ο κύριος Λάγκε. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Πολλά και σωστά επιχειρήματα ακούστηκαν. Το πρώτο είναι νομική βάση. Η νομική βάση προτείνει να επιφορτιστεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να επιφορτιστεί με αυτό. Στο άρθρο 127.6 αναφέρεται αυτό ρητός, αλλά επίσης ρητός η εξαίρεση των ασφαλιστικών εταιριών. Αλλά δεν είναι ε, αμυγός ε, παρκές αυτό το επιχείρημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Δεν είναι τόσο απλό. Ε, δεύτερο, το γεγονός ότι το έπραξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί να αντιδράσουμε. Διότι οι επιφυλάξεις ακούστηκαν και είναι πολλές. Σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ τραπεζικής εποπτείας και νομισματικής πολιτικής. Κεντρικές τράπεζες και ε, εποπτεία τραπεζών αμειγνύονται, οπότε ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος. Ε, η ε, δημοκρατική νομιμότητα εκφράστηκε. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα μέλος του Διευθυντηρίου της ΕΚΤ που είναι αρμόδια για την νομισματική πολιτική στο μέλλον να είναι αρμόδιο για την εποπτεία των τραπεζών. Όχι, θα πρέπει να είναι τελείως ανεξάρτητο από τις υφιστάμενες δομές στο σύστημα, ξεχωριστό. Κάτι άλλο που προτείνω εγώ για το δημοκρατικό έλεγχο δεν αρκεί να μας ακούνε ή να λογοδοτούν σε εμά, δεν είναι απλή ακρόαση σύμβουλη, αλλά όπως συμβαίνει και στη Γερμανία, στην Πάφιν, ε, στην εποπτεία των τραπεζών θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις ευρωβουλευτές στο εποπτικό συμβούλιο. Και ε, από τους τρεις μία τουλάχιστον να είναι γυναίκα, τουλάχιστον. Και πιστεύω ότι επικεφαλής επίσης θα πρέπει να εκλέγεται από το Κοινοβούλιο και όχι απλώς να αλαμβάνει γνώση το Κοινοβούλιο γι' αυτό. Το χρονικό επίσης πλαίσιο είναι τελείως ανεπαρκές. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτή τη στιγμή έχει 57 υπαλλήλους, είναι πάρα πολύ αξιόλογοι και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά στα κράτη-μέλη έχουμε εποπτικές αρχές για ασφάλειες ε, χρηματιστήρια και τράπεζες και εκεί εργάζονται 53.000 άνθρωποι στην Ένωση, 53.000. Και θα ήταν πάρα πολύ λάθος να πούμε ότι ε, μεταφέρουμε αυτές τις αρμοδιότητες τις σημαντικές για τις τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χωρίς να έχουμε εξηγήσει το διαχωρισμό και το πλαίσιο των καθηκόντων και χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε αυτό το δυναμικό. Και σε αντίθεση με κάποιους συναδέλφους, πρέπει να πω ότι στο άρθρο 127.6 αυτά που λένε για την ΕΚΤ θα πρέπει επιπλέον να έχει υποπροζώνη Είναι γελία αυτά που προτείνονται στον κανονισμό για την τραπεζική αρχή. Εκεί λέει η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πώς θα έχει. Η Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή μπορεί να συντονίζει και να προσκαλείται ως παρατηρητής. Τι είναι αυτό. Ευνοχισμός καταργούμε την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, ε, την ε, κάνουμε κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εάν θέλουμε να διαπραγματευτούμε μαζί, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να περιοριστεί στα όσα προβλέπονται από τις συνθήκες και να πιέσουμε ε, σε μια ενιαία αγορά να έχει τη βασική αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Εμείς αγωνιστήκαμε γι' αυτό και τώρα έρχονται και το καταργούν τι να την κάνουμε την ενία ε, τραπεζική εποπτεία αν στο τέλος 60% ε, των τραπεζών, 60% των χρηματαγορών, των χρηματοπιστωτικών Μεγάλη Βρετανία ε, βγαίνει απ' έξω. 60% το επαναλαμβάνω. Πού είναι η ενιαία εποπτεία. Το αντίθετο επιτυγχάνουμε. Διχοτόμηση της Ευρώπης με μεγάλη εκρηκτική κατάσταση και κινδύνους και θα ήθελα να ε, πω τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη σελίδα 2 για τον κανονισμό. Ε, στη Σύνοδο Κορυφή των, ε, της Ευρωζώνης, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ζητούν σύντομα να κάνει προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για νέο μηχανισμό. Μόλις δημιουργηθεί ένα τέτοιο σύστημα για την ΟΝΕ, μετά από μια σωστή απόφαση θα έχει τη δυνατότητα άμεση ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό σταθερότητα. Α, σε αυτό αποσκοπεί λοιπόν για την Ισπανία κυρίως άμεση ανακεφαλαιοποίηση των ε, τραπεζών στην Ισπανία διότι δεν θέλει η Ισπανία να μπει στο μνημόνιο να κάνει τέτοια αίτηση. Και έτσι όμως με αυτό τον παράδρομο και την παράκαμψη όχι μόνο παραβιάζεται η συνθήκη, αλλά ε, διακυβεύεται και αφισβητείται και ολόκληρο το σύστημα εποπτείας των τραπεζών στην Ευρώπη. Και η ΕΚΤ αύριο δηλαδή θα πρέπει να ελέγχει 6.200 τράπεζες στην Ένωση και μικρές περιφερειακές τράπεζες, τοπικές αυτό είναι τελείως απαράδεκτο. Θα πρέπει να παραμένει αυτό εθνική αρμοδιότητα. Και είμαι βέβαιος ότι θα φροντίσει η Μεγάλη Βρετανία να γίνει αυτό. Γιατί η απόφαση βάσει το άρθρο 127.6 θα πρέπει να είναι ομόφωνη. Ομόφωνη ίσον ε, του κοινό παρανομαστής, μέγιστο δυναμικό εκβιασμού, ερήμην του Κοινοβουλίου και δεν συμφωνώ καθόλου. να δώσουμε αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να συνδεθεί με το μηχανισμό σταθερότητας. Αυτό είναι δικαιολογημένο και θεμητό όπως ζητάει η Ισπανία. Αλλά ενιαίος ευρωπαϊκός μηχανισμός ε, εποπτείας να μπει στην ΕΜΠΑ, στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και όχι στην ΕΚΤ. Και όχι άρον-άρον να τρέχουμε. Ε, δεν θέλουμε, διαφωνούμε με την πρόταση αυτή. Και δεν φταίμε εμεί ε, για την πίεση χρόνου, ούτε γεννήθηκε από την κρίση αυτό. Απλώ μόνο επειδή ισχυρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η Dexia, η Bankia, η Northern ε, Rock ε, είναι μικρές τράπεζες. Δέξια 511 δισεκατομμύρια το 10 ε, πριν δημιουργηθεί η Bad Bank. Ο εισαγωγισμός, η, η Bankia στην Ισπανία 311 ε, δις τζίρο, το 2006 Northern Rock πριν να βαγίσει 150 δις. Δεν είναι μικρές περιφερειακές τράπεζες. 70 δις έχουμε, από τα 70 δις ε, ισολογισμό και πάνω ε, θεωρείται μεγάλη μια τράπεζα. Και εάν τα συμπληρώσουμε αυτά και με κάποιε άλλε δηλώσει του κυρίου Ντράγκη σε κεκλεισμένο των θυρών συνεδρίαση ότι πρέπει να βρεθεί ένα τρόπο, μία ε, φόρμουλα να υπολογίζονται αυτά, τότε μπορούμε να κατέβουμε και κάτω από τα 70 δις, εάν πληρούν αυτές τις τρεις προϋποθέσεις οι τράπεζες. Και αυτό θα ήταν ε, η εφετηρία για μια εποπτεία που ε, θα είναι ενιαία και δεν θα διακυβεύει ούτε την ΕΜΠΑ ούτε τις Εθνικές Εποπτικές Αρχές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λάγκεν. Τι να κάνω να συνεχίσουμε τώρα αυτή τη συνεδρίαση δηλαδή. Γκούνερ Χόκμαρκ, σας ευχαριστώ πολύ και είμαι ευτυχής γιατί μπορώ να συμφωνήσω με πολλά από όσα υπόθηκαν σήμερα το πρωί ήταν πολύ σημαντικές σκέψεις και προβληματισμοί. Θα πρέπει νομίζω να διαπιστώσουμε το κίνδυνο που διατρέχουμε να διχάσουμε την Ένωση και να την καταστήσουμε πιο αδύναμη. Ενώ επιθυμούμε το, το αντίθετο. Για, γι' αυτό το λέω ότι γιατί ακόμα και αν φτιάχνουμε μια δομή για ε, σωστούς λόγους, ε, συνήθως ε, αποκτά δική τη ζωή μετά ο κάθε οργανισμός και ενεργεί πιο αυτόνομα. Και αυτό θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε κίνδυνο κατακαιρματισμό όχι μόνο για τις <laughs> δημοσιονομικές αγορές όσον αφορά τους κανόνες, πώς εφαρμόζονται αυτοί, αλλά και κατακαιρματισμό της ίδιας της ενιαίας αγοράς. Διότι όταν ξεκινά ένα πολιτικό σώμα, όταν ξεκινά μια τέτοια διαδικασία, μπορεί να συνεχιστεί επάπειρον. Αλλά θα ήθελα επίσης να πω, και αυτό συνάδει με τα όσα είπε ο κύριος Λάγκε, ότι πιστεύω πως είναι εύκολο να δούμε και να καταλάβουμε πως χρειαζόμαστε καλύτερη εποπτεία. Όταν όμως ακούμε κάποιες από τις παρεμβάσεις εδώ σήμερα και ακόμα περισσότερο όταν βλέπουμε κάποιες προτάσεις που, ακούσα, που υπήρξαν, που έγιναν, ε, είναι σαν να αγνοούμε το γεγονός, και εδώ θα σας αποκαλύψω και ένα μυστικό, πως ήδη υπάρχει εποπτεία δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι την έχουμε σε εθνικό επίπεδο και την έχουμε και μέσω μιας νομοθεσίας την οποία ολοκληρώσαμε πριν από ένα χρόνο νομίζω μόνο. Ακριβώς. Δηλαδή μην λέμε για την εποπτεία, λες και είναι κάτι το ανύπαρκτο και το οποίο πρέπει να φτιάξουμε από την αρχή. Απλώς θέλουμε να φτιάξουμε μια εποπτεία που ελπίζουμε ότι θα είναι καλύτερη από αυτή που ήδη έχουμε. Και αυτό όχι μόνο επειδή κινούμεθα ή δημιουργούμε μια νέα, ένα νέο οργανισμό, αυτό είναι σημαντικό να το κάνουμε. Δηλαδή, εφόσον φτιάχνουμε μια δομή για την εποπτεία, που από τη φύση της αποκλείει το ίμιση των ε, δημοσιονομικών αγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου οι αγορές είναι εξαιρετικά ολοκληρωμένες, τότε μπορεί να δημιουργήσουμε περισσότερους κινδύνους και προβλήματα από αυτά που προσπαθούμε να επιλύσουμε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, κύριε Πρόεδρε. Στις σκανδιναβικές χώρες είναι πολύ ολοκληρωμένες οι τράπεζες. Σουηδία, Δανία, Φιλανδία, Νορβηγία, Εστονία. Λετωνία και Λιθουανία. Τραπεζικό τομέα, ε, μάλλον ασφαλίσεις και χρηματιστήρια. Πολύ, ε, πολύ κλειστό κύκλωμα. Δίκτυο. Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε τώρα μια εποπτική δομή που θα αποκλείει το μισό όλων αυτών. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν σοφό. Αυτό που λέω εγώ δεν είναι επιχείρημα κατά Τη δημιουργίας μια ισχυρότερη εποπτείας ανάμεσα στα κάποια κράτη-μέλη. Αυτό που λέω είναι ότι δεν πρέπει να δεχτούμε να αναπτύξουμε μια δομή που, δίνει, που κάνει κάποιο είδους διατησίες για όσου θέλουν να ξεφύγουν από πιο έντονη εποπτεία. Βασικός μας στόχος βέβαια θα πρέπει να είναι να εξασφαλίσουμε πω η εθνική εποπτεία λειτουργεί και ότι έχουμε κοινά ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που μπορούν αυτά να τα παρακολουθήσουν με διάφορους τρόπους, αλλά να μην πιστεύουμε <clears throat> ότι θα επιτύχουμε καλύτερη υποπτή από αυτή που ήδη έχουμε. Σήμερα είμαστε 27, 27 εθνικές αρχές και η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και οι άλλες αρχές που έχουμε. Πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι όλα αυτά θα λειτουργήσουν καλύτερα. Θα γίνουν καλύτερα και αν θέλουμε να αναθέσουμε κάτι στην ΕΚΤ που μπορεί να αμφισβητηθεί γιατί έτσι θα δώσουμε διπλή έργο στην, στην ε, ΕΚΤ. Να δούμε όμως αν όλα αυτά είναι αξιόπιστα, να μην χάσουμε τη γενικότερη ευκαιρία που έχουμε για να ενισχύσουμε την μέσω και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Απλώς λοιπόν επειδή εφευρίσκουμε μια νέα αρχή, μια νέα δομή, δεν σημαίνει πως την φτιάχνουμε και καλύτερη. Πρέπει σε αυτή να βασιστούμε και να οικοδομήσουμε βήμα προς βήμα. Και νομίζω πως αυτό είπαμε όλοι, αριστερά και δεξιά σε αυτήν την Επιτροπή και είναι καλή κοινή ε, αρχή για τις μελλοντικέ μας εργασίες. Ευχαριστώ. Η κυρία Ελίζα Φερέιρα. <laughs> Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω πως ε, γίνεται εδώ μια συζήτηση που είναι εξαιρετικά σημαντική. Και ε, θα ήθελα πέρα από τα όσα ήδη υπόθηκαν να υπογραμμίσω ε, δύο-τρία δύο, σημεία. Εν γέννη, εμείς υποστηρίζουμε έναν ε, μοναδικό, έναν ενιαίο επόπτη για ολόκληρη την Ευρώπη και, την, ε, ε, και αυτό ήδη από τον Ιούνιο του 2010. Εν τω μεταξύ υπήρξαν πολλές πρωτοβουλίες που, αλλά μόνο τώρα έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις από πλευράς της Κομισιόν. Και Πρέπει να υπάρχει συνοχή ανάμεσα σε όλες αυτές τις ε, προτάσεις και το Κοινοβούλιο πρέπει να προσέξει. Καταρχήν αυτά που είπε ο κύριος Χόκμαρκ όσον αφορά την ε, ε, εξαγορά, εξυγίανση τραπεζών και τις αρμοδιότητες της ΕΚΤ και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής στο πλαίσιο της Τραπεζικής Ένωσης. Όταν ε, τότε έλαβε θέση το Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα, σκεφτόμα, δίναμε μια πολύ μεγάλη εξουσία στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή που θα είχε βασικό ρόλο για τα συστημικά ε, θεσμικά όργανα και για την εποπτεία αλλά και για περιπτώσεις πτώχευσης. Αυτή τη εγώ θα πρέπει να αναγνωρίσω και οφείλω να αναγνωρίσω ότι η πρόταση που αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή της λειτουργίας της εποπτείας στην Ευρωζώνη ε, να έχει αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα τουλάχιστον σε δύο επίπεδο. Από τη μια πλευρά έχει δυνατότητα να παρέμβει, ε, είναι ισχυρό αυτό το θεσμικό όργανο και είναι ε, και αξιόπιστο και έχει ένα κύρος, σε πάση περιπτώσει. Τώρα θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιηθεί αυτό το κύρος. Φυσικά και είμαι πολύ ευαίσθητη όσον αφορά τα θέματα της συνοχής ανάμεσα στις πρακτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ε, των υπολείπων εποπτών. Ε, θα έλεγα λοιπόν ότι ένας πιθανός δρόμος είναι η εναρμόνιση, η πιο γρήγορη εναρμόνιση πρακτικών εποπτείας μέσω και έξω από τη ζώνη ευρώ. Αυτό αν δεν θέλουμε να θέσουμε σε κίνδυνο τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Δεύτερη παρατήρηση ότι αυτή η συνοχή θα πρέπει να είναι εγγυημένη και μέσα στην ευρωζώνη, έτσι ώστε το να έχουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να απορροφήσει ως μοναδικός επόπτης ε, τις εθνικές πρακτικές ε, εποπτείες και εκεί θα πρέπει να συνεχίσουμε και να, να ζητάμε από την έκτη να αναγνωρίσει τα όργανα εθνικής εποπτείας ως πολύ σημαντικά στοιχεία στην οικοδόμηση μιας κοινής κουλτούρας εποπτείας εντός της Ένωσης. Εδώ φυσικά υπάρχει και το θέμα της σχέσης ανάμεσα στις τράπεζες και στην εποπτεία των τραπεζών, αλλά και στην εποπτεία των ασφαλιστικών εταιριών, αλλά και με το παράλληλο τραπεζικό σύστημα, όπου και εκεί θα πρέπει να λυθεί το θέμα και να αποφασίσουμε και είχα την ευκαιρία να θέσω την ερώτηση στην συνεδρίαση που κάναμε την περασμένη εβδομάδα ε, πώς γίνεται να μην έχουμε σκεφτεί την εποπτεία των ομίλων ε, και των ασφαλιστικών εταιριών. Ε, πρέπει πραγματικά να δουλέψουμε για την πραγματική και γνήσια ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας, γιατί όταν η Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να αποφασίσει για τις τράπεζες και για το μέλλον των τραπεζών που έχουν, ε, που έχουν ε, μεγάλη κάλυψη πολλές χώρες θα υπάρχουν πολλά ζητήματα Ποιο, και θα πρέπει να σκεφτούμε επίσης ποιον μηχανισμό έφεσης δυνατότητας προσφυγής θα έχει η τράπεζα αυτή όταν στην άσκηση της εποπτείας ε, θίγονται εθνικά συμφέροντα και πώς θα γίνει η μετάβαση από αυτή την εποπτεία που συμπεριλαμβάνει αυτό που ονομάζεται early intervention, έγκαιρη παρέμβαση για την ε, ε, εξαγορά των τραπεζών, την εξυγίαση των τραπεζών, ώστε ε, να περάσουμε στην επόμενη φάση όπου μια τράπεζα κάνει πτώχευση, πράγμα το οποίο έχει επιπτώσεις όσον αφορά τον προϋπολογισμό και που επιπτώσεις οι οποίες δεν έχουν ε, ληφθεί υπόψη. Αυτό είναι το θέμα της ΕΚΤ σε περιπτώσεις ε, της Ευρωζώνης και σε περιπτώσεις τραπεζών που λειτουργούν σε διάφορες χώρες θα πρέπει να δει τα σχέδια εξυγίανσης της τράπεζας αλλά η πραγματική πώληση της τράπεζας, η εξαγορά αυτής, θα πρέπει να γίνει από την εθνική, από το εθνικό επίπεδο, όχι από την εγκεντρική τράπεζα. Και αυτά θα πρέπει πολύ καλά να το δουλέψουμε. Να υπάρχει μία ενιαία εποπτεία, αλλά και μια δύσκολα θα γίνει εάν δεν υπάρχει και ένα ταμείο εξυγίανσης και μια αρχή ε, εξυγίανσης ή εξαγοράς των τραπεζών. Θα πρέπει δηλαδή η αρχαία η εποπτική να έχει και αρκετό βάρος όσον αφορά την παρέμβασή της. Και εδώ έρχεται ο ρόλος της ε, EBA που θα πρέπει να παίξει τεράστιο ρόλο όσον αφορά τη δημιουργία μιας κοινή ε, κουλτούρας για την εξαγορά ή την εξυγίανση των τραπεζών και θα πρέπει αυτό το θέμα να το εξετάσουμε εις βάθος. Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να λάβουμε κάποια συγκεκριμένη θέση όσον αφορά την προσαρμογή ε, με βάση τα όσα θα γίνονται. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε την επόμενη εβδομάδα να εξετάσουμε την έκθεση Λικάινεν. Θα υπάρξουν εξελίξεις επίσης τον Οκτώβριο και άλλες φάσεις ε, ε, για την Τραπεζική Ένωση. Και άρα λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσουμε τη στρατηγική μας ως Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα όσα πρέπει να αποφασιστούν σε πολιτικό επίπεδο. Να έχουμε λοιπόν από τη μια πλευρά τις πολιτικές μας και από την άλλη να έχουμε και μια δραστήρια παρουσία. Να μην περιμένουμε δηλαδή μέχρι το τέλος των διαδικασιών ενώ το πλαίσιο αλλάζει στην πορεία. Έχουμε κάνει σημαντική δουλειά μέχρι στιγμή στο Κοινοβούλιο, αλλά πιστεύω πως θα πρέπει να προχωρήσουμε με πολύ δραστήριο τρόπο, ενεργά, για να συμμετέχουμε δραστήρια σε αυτή τη διαδικασία και να πετύχουμε τους στόχους μας και να μην ξεχνάμε ότι η κατάσταση από την οποία ξεκινάμε δεν λειτουργήσε. Δυσώθηκαν οι τράπεζες από τους φορολογούμενους και υπάρχουν τράπεζες που είναι πιο ισχυρές από ότι οι χώρες που τους φιλοξενούν. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν λέγοντας ότι μικροβελτιώσεις και μικροαυξήσεις στην κατάσταση μπορεί να βελτιώσουν ε, τα πράγματα. Δεν πρόκειται να γίνει γίνει κάτι τέτοιο. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει, ε, μάλλον πιστεύω ότι θα πρέπει να καλύψουμε το πολιτικό χώρο που μας έχει ανοιχθεί με ε, τα κατάλληλα βήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Now, uh, please, Mrs. Intveld. Ευχαριστώ κύριε Νετβέλ voorzitter. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Dat de discussie wel duidelijk maakt. Ε, τι φαίνεται από τη συζήτηση, ότι έχουμε ένα δίλημα εδώ. Από τη μια, θέλουμε μια γρήγορη λύση. Εξού και η ΕΚΤ, ο καθένας αναγνωρίζει ότι ε, υπάρχουν ε, διαμαρτυρίες, γιατί η λύση που δίνεται δεν είναι επαρκής. Οπότε, Τώρα, υπό τη χρονική αυτή πίεση θα πρέπει να επιλέξουμε ε, κάτι το οποίο θα ισχύσει διαπαντός. Ε, εμείς δεν μπορούμε να βρούμε κάποια ενδιάμεση λύση. Ε, έτσι, κάτι βράχει πρόθεσμο ε, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που είναι η μόνη ρεαλιστική, εν πάση περιπτώσει, πρόταση. Βράχει πρόθεσμα, επαναλαμβάνω. Αλλά να πούμε ότι θέλουμε λίγο χρόνο για να συζητήσουμε και να καταλήξουμε στην οριστική πρόταση για την εποπτεία που έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Παράδειγμα, θα μπορούσα να φανταστώ να πούμε ότι προς το παρόν να μπει αυτό στην ΕΛΚ, ΕΚΤ με τρόπο πάρα πολύ ξεχωριστό, εντάξει, ε, και τελικά ε, να μπει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, μια άλλη δομή εποπτείας ε, στο απότερο μέλλον. Δεν ξέρω τεχνικά αν γίνεται αυτό και από πλευρά συνθήκων. Ε, πάντως εγώ δυσκολεύομαι τώρα άρον άρον να πιεστούμε, να βρούμε μια λύση οριστική και αμετάκλητη και μετά να μην μπορούμε να την ε, αλλάξουμε. Να πούμε ότι θέλουμε χρόνο αλλά δεν υπάρχει καμία ε, εγγύηση ότι θα φτάσουμε ε, στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Οπότε αυτό θα ήθελα να ζητήσω, να εξετάσουμε αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Να ε, επιλέξουμε τώρα μια ενδιάμεση λύση, βράχη πρόθεσμα για να λύσουμε αυτό το θέμα, αλλά πιο μακροπρόθεσμα με την ησυχία μας να σκεφτούμε τι θέλουμε ακριβώς και πώς θα το διαμορφώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Βότμαν Κόλ. Πολλά ακούστηκαν μέχρι τώρα και με τα οποία συμφωνώ να υπογραμμίσω όμως τρία βασικά θέματα. Πρώτον, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμήσουμε την ανάγκη να προχωρήσουμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το ενιαίο εποπτικό πιστοτικό σύστημα στην Ευρώπη, γιατί όχι μόνο έχουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα του υπερβολικού δημοσίου χρέους, αλλά έχουμε ένα θέμα εμπιστοσύνης στο πιστοτικό μας σύστημα και αυτό είναι κάτι το οποίο ξεπερνά τα τοπικά προβλήματα όπως αυτά που αντιμετωπίσαμε εδώ με τον Τέξια. Οι νομικές αξιολογήσεις τις οποίες διάβασα νομίζω ότι δεν δίνουν την δυνατότητα να αφισβητήσουμε την οδική βάση την οποία χρησιμοποιεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το θέμα είναι ότι οι προτάσεις αυτές δεν έχουν οριμάσει ακόμα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν να αντιμετωπιστούν σαν πακέτο. Η εμπλοκή του Κοινοβουλίου και στα δύο αυτά θέματα θα πρέπει να υπάρξει όπως και στην περίπτωση του εξαπλού πακέτου. Τότε είχαμε τέσσερις προτάσεις επί τη βάση των προτάσεων, επί τη βάση της συνθήκης μάλλον και το Συμβούλιο τις αντιμετώπισε με ισότιμο και ενιαίο τρόπο. Περιμένω λοιπόν από τους εισηγητές μας να μου πούν αν κάτι τέτοιο το έχει αναγνωρίσει η Επιτροπή και το Συμβούλιο. Από το Συμβούλιο είδα κάποια, από την Επιτροπή μάλλον είδα κάποια μηνύματα. Ο πρόεδρος Μπαρόσο είπε ότι οι προτάσεις αυτές συνδέονται μεταξύ τους και θα τις προωθήσει ενιαία. Σχετικά τώρα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η διαφορά ανάμεσα στην ανεξαρτησία την οποία έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στον τομέα το νομισματικό και στο νέο αυτό τον εποπτικό τομέα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει νομικά πιο βέβαιο, πιο ασφαλές και το θέμα του ελέγχου και του υπολόγου σε εισαγωγικά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ισχύσει και στην περίπτωση της ενίας εποπτικής αρχής. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να υπάρξει εμβάθυνση και σε σχέση με τον αριθμό των πιστοτικών ιδρυμάτων και σε σχέση με τον αριθμό των χωρών που θα πάρουν μέρος. Γι' αυτό απαιτείται κάποιος χρόνος βέβαια. Το βασικό είναι να διευκρινίσουμε ότι το σύστημα θα πρέπει να ισχύσει για όλες τις χώρες ή εν πάση περιπτώσει για όσες περισσότερες γίνεται και πρέπει να προκαλέσουμε τις χώρες να πάρουν μέρος. Και σαφώς αυτό θα πρέπει να επεκταθεί ε, σε όλες τις τράπεζες. Βέβαια αυτό που μας ενδιαφέρει χρονικά είναι οι λεγόμενες συστημικές τράπεζες, οι μεγάλες, αλλά και για τις μικρές τράπεζες θα πρέπει να υπάρξει ένα ενιαίο σύστημα. Βασική μου ανησυχία είναι ότι όταν βλέπει κανείς αυτές τις δύο προτάσεις, στην ουσία υπονομεύουν κάποιες θέσεις οι οποίες ακούστηκαν σχετικά με την Ευρωπαϊκή ε, Τράπεζα, είναι, ε, την EBA μάλλον, την Εποπτική Αρχή την πιστοτική εποπτική αρχή. Είναι αλήθεια ότι δεν θα πρέπει να υπονομεύσουμε την εποπτική αρχή, ιδιαίτερα στα πεδία στα οποία είναι ήδη υπεύθυνοι. Γιατί όταν μιλάμε εμείς ε, ότι θα πρέπει να έχουν τη διακριτική ευχέρεια οι εθνικές εποπτικές αρχές να ελέγχουν την κατάσταση, αυτή ακριβώς την ευχέρεια θα πρέπει να τη μεταφέρουμε εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η διατήρηση της ενιαίας αγοράς πρέπει να είναι βασικός στόχος μας. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να φύξουμε. Συμφωνώ και με τους προλαλήσαντες οι οποίοι ζήτησαν χρόνο. Βέβαια θα συμφωνήσω ότι η ποιότητα προηγείται της ταχύτητας. Από την άλλη όμως, διατηρώντας την ποιότητα μπορούμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες για να μην καθυστερούμε άλλο, γιατί τα προβλήματα στην Ευρώπη σήμερα τα οικονομικά είναι σοβαρότατα <laughs> και πρέπει να πάρουμε κάποια αξιόπιστα, να κάνουμε κάποια αξιόπιστα πρώτα βήματα. Ευχαριστώ, λέει ο Ο κύριος Νταφ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε, προέρχομαι από μια άλλη ε, κοινοβουλευτική επιτροπή και σας μεταφέρω τους αδελφικούς χαιρετισμού της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Σας μεταφέρω επίσης και μια προειδοποίηση. Νομίζω ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως έχουν δημιουργούν σοβαρότατα προβλήματα στην οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βασικό πρόβλημα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα προσπαθήσουμε η εποπτική αυτή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να ε, λειτουργήσει με διαφάνεια, με έλεγχο ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει η τράπεζα να διατηρήσει την ανεξαρτησία της ή τουλάχιστον αυτό της έχουμε υποσχεθεί. Υπάρχουν εδώ και πολιτικές πλευρές τις οποίες θα πρέπει να εξετάσουμε, αλλά και νομικές βέβαια. Tyson ought in, uh, uh, to try to η κυρία Τίσεν προσπάθησε ακριβώς να μας μεταφέρει θα έλεγα αυτό το συνικό τείχος το οποίο έχει αρχίσει και περιβάλλει πλέον τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και τίθεται φυσικά και το θέμα του δημοκρατικού ελέγχου της, του οργανισμού αυτού, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά από και τα, από και τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι δεν υπάρχουν δύο κατηγορίες κρατών μελών, αλλά τρεις. Είναι αυτές που είναι μέσα στην ε, Ευρωζώνη, είναι αυτές που είναι έτοιμες να μπουν στην Ευρωζώνη και ανάμεσα σε αυτές που είναι έτοιμες να μπουν στην Ευρωζώνη υπάρχουν χώρες που έχουν ανεξάρτητο πιστοτικό τομέα με ανεξάρτητη εποπτεία και άλλες που έχουν κεντρικά ελεγχόμενο. Και η τρίτη, η τρίτη κατηγορία είναι οι χώρες οι οποίες ε, θέλουν να μείνουν εκτός και εδώ τίθεται το θέμα βέβαια γιατί ανάμεσα σε αυτές τις χώρες είναι το Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο έχει το μεγαλύτερο ποσοστό των πιστοτικών δραστηριοτήτων κτλ. Λοιπόν, ένα πρώτο συμπέρασμά μου είναι ότι θα πρέπει να οδηγηθούμε σε μια εναλλακτική ριζοσπαστική λύση, την δημιουργία δηλαδή ενός πραγματικά ενιαίου χώρου όλοι να παίζουν στην ομάδα. Μία αρχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ευρωπαϊκή η οποία θα αντικαταστήσει ουσιαστικά τις εθνικές εποπτικές αρχές. Αυτή είναι μια επιλογή την οποία αν μη τι άλλο θα πρέπει να τολμήσουμε να συζητήσουμε πριν να περάσουμε στην αποδοχή της νομικής βάσης η οποία προτείνεται από πλευράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με το σύστημα το εποπτικό το οποίο θα πρέπει γρήγορα να τεθεί σε λειτουργία. Και μια τελική σκέψη, βασισμένη στις εμπειρίες που είχαμε μέχρι σήμερα. Το Συμβούλιο Υπουργών είναι πάρα πολύ πιθανό να τα κάνει σαλάτα για μια ακόμη φορά. Σε ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Κάρινς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχουν υποθεί πάρα πολλά. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, όπως πάντα άλλωστε. Ποιος είναι ο δικός μας ρόλος να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εσωτερική αγορά. Και όταν μιλούμε για την τραπεζική εποπτεία ή απλώς την τραπεζική ένωση, θα πρέπει να αναρωτηθούμε οι αποφάσεις που θα λάβουμε θα ενισχύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ή μήπως θα την αποδυναμώσουν, όπως είπε ο Γκούναρ, γιατί θα τη διχάσουν ενδεχομένω. Στην Ευρώπη έχουμε διαφορετικό είδος αγορών, ε, μάλλον εμπιστοσύνη ε, της αγοράς. Οι αγορές δεν ε, εμπιστεύονται πάντα τα θεσμικά όργανα και έχουμε και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Αν τα κάνουμε στραβά, τελικά όχι μόνο θα, δεν θα επανέλθει η εμπιστοσύνη των αγορών, αλλά θα διαλυθεί και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, που μέχρι σήμερα δεν υπάρχει παντού. Στη χώρα μου, τη Λετωνία, λήφθη μια απόφαση, ε, μάλλον ε, το φθινόπωρο του 2008 έλαβε μια απόφαση η Ιρλανδία για να καλύψει όλες τις ε, καταθέσεις με εγγυήσεις χωρίς καμία εξαίρεση. Και αυτό είχε επιπτώσεις και στη χώρα μου, τη Λετωνία και παντού, γιατί ε, το 70% των ε, τραπεζών ε, των δικών μας ήταν σκανδιναβικές, που είναι βέβαια εκτός ευρωζώνης, αλλά ορισμένες ήταν και εντός και το 30% ήταν λετονικές. Και αφού αποφάσισαν οι Ιρλανδοί να καλύψουν όλες τις καταθέσεις, το αποφάσισαν και οι Σουηδοί και για τις τράπεζές τους και τις θηγατρικές. Και εκεί έτρεξε ο κόσμος να πάρει τις κατεθέσεις του και αυτό ε, και να αλλάξει τράπεζα ε, κόστισε ένα δισεκατομμύριο στους φορολογούμενους και η χώρα μου δεν το είχε ούτε τα δύο δις ε, απευθύνθηκε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για διάσωση και τα γνωστά. Ε, καταλαβαίνετε λοιπόν, μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πήρε μία απόφαση ε, και ε, χωρίς να αποσκοπεί σε αυτό είχε πάρα πολύ αρνητικές ε, επιπτώσεις και διακλαδώσεις αυτή η απόφαση σε άλλες χώρες της Ένωσης. Λοιπόν, όταν συζητούμε για εποπτεία των τραπεζών θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί να μην διευρύνουμε ακόμα περισσότερο κάποια χάσματα που υπάρχουν ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν υπάρχει λοιπόν μια τέτοια αρχή Κεντρικέ λοιπόν εξουσίες ενισχυμένες, θα πρέπει αυτό να καλύπτει το σύνολο τη Ένωση. και την Ευρωζώνη και εκτό Ευρωζώνη και γενικότερα. Κανονικά θα πρέπει να καλύπτει όλα τα κράτη-μέλη. Για φανταστείτε μια κατάσταση σαν την Εστονία που είναι σήμερα στην Ευρωζώνη. Αλλά οι τράπεζε της είναι ξενε από χώρε εκτό Ευρωζώνη. Αυτό πώς θα γίνει τώρα, πώς θα λειτουργήσει το σύστημα. Οι εστονικές τράπεζες πώς θα καλύπτονται. Με το Ηνωμένο Βασίλειο τι γίνεται που είναι εκτός και ήδη σου λένε προς Θεού δεν θα μπούμε ποτέ. Αλλά ε, υπάρχουν τράπεζες στη Μεγάλη Βρετανία που λειτουργούν και είναι τράπεζες της Ευρωζώνης. Πώς θα γίνει η εποπτεία πανευρωπαϊκά. Να μην ενισχυθεί η διαίρεση αντί να ενισχυθεί η εποπτεία. Όχι μόνο θα επικρατεί ασάφεια στις αγορές, αλλά τι γίνεται με τους καταναλωτές. Και ε, θα έχουμε ροέ κεφαλαίων, θα φεύγουν από τη μια χώρα στην άλλη, από τη μια τράπεζα στην άλλη, με τελείω χαόδη τρόπο, ε, επιβλαβή για όλου. Λοιπόν, αν γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι πάντε και να δούμε πώ μπορεί να γίνει αυτό, αν είναι στην ΕΚΤ με τα νομικά εμπόδια και περιορισμού. τι θα γίνει με τα δικαιώματα ψήφου και αντιπροσώπευση κρατών εκτό τη Ευρωζώνη. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε, να τα απαντήσουμε και να ληφθούν υπόψη. Δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα ποτέ δεν ήταν εύκολο, έτσι δεν είναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η Ρουμανία δεν είναι στην Ευρωζώνη, αλλά έχει τράπεζες ε, από την Ευρωζώνη που λειτουργούν στη Ρουμανία. Μάλιστα. Ο κύριος ε, Νίκλας. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, Πρόεδρε. Και να αντιδράσω στα όσα είπε ο κύριος Κάριντς που είπε ότι το 70% των τραπεζών στη χώρα του ήταν σε ξένα χέρια. Στην Πολωνία η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη, μόνο το 60% είναι ξένες τράπεζες. Η νέα αγορά είναι πολύ ωραία, πολύ καλό πράγμα. Αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας τα εξή. Στην Πολωνία έχουμε πολλές ισπανικές τράπεζες. Το εγχώριο μας τραπεζικό σύστημα δεν αποτελείται από αδύναμες τράπεζες. Έχουμε καλές τράπεζες. και ε, γίνονται συζητήσεις, μάλιστα ορισμένες έχουν ολοκληρωθεί επιδιχώς, για να εξαγορά των ισπανικών τραπεζών από τις πολωνικές. Όμως αυτή η διαδικασία διεκόπη λόγω του ερωτηματικού αυτού για την τραπεζική εποπτεία στην Ισπανία για τις, ε, την πιθανή μελλοντική ανακεφαλοποίηση των Ισπανικών τραπεζών. Ακόμα και σήμερα λοιπόν η ενιαία αγορά δεν λειτουργεί σωστά στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε διαφορετική κατάσταση από το Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο έχει το opt-out. Εμείς ε, οδεύουμε προς την Ευρωζώνη. Η πολωνική κυβέρνηση είπε πως η Πολωνία θα έμπαινε στην Ευρωζώνη το 2012. Εντάξει, ήταν λίγο όνειρα, τρελά αυτό, αλλά ε, εν ο στόχος μας είναι η Ευρωζώνη. Mm. Είμαι βέβαιος πως όλοι είδατε σήμερα το πρωί τις εικόνες από τη Μαδρίτη. Αλλά το γεγονό είναι ότι οι πιο ενθουσιώδης ε, υπέρ του ευρώ είναι αυτοί που δεν είναι στο ευρώ. Mm. Όπως η Πολωνία. Και δεν νομίζω θα πρέπει αυτό να το αγνοήσουμε το θέμα, όπως ε, το κάνει και η Κομισιόν στο έγγραφό της. Και να πω και κάτι ακόμα. Για αρκετές χώρες... Είναι αυτό προφανέ. Εμείς στην Πολωνία, να πω κάτι ακόμα, προχωρούμε ναι, με φουλ ταχύτητα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Και δεν ήταν πάντοτε ομαλά τα πράγματα. Ε, δεν είμαστε πλήρη, πλήρη μέλη της ενιαίας αγοράς. Έχουμε ταλαιπωρηθεί για 7 χρόνια μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία απαγόρευσαν ε, στον λαό μας να δουλεύει στην επικράτειά τους. Και τώρα χώρες όπως η Πολωνία που πέρασαν αυτή την ε, περίοδο σνομπαρίσματος και δεν θέλω τώρα εγώ να αρχίσω να τα βγάζω στη φόρα, αλλά υπάρχουν κάποιες χώρες, κάποιες χώρες που θέλουν να ανακατευτούν στην πολωνική εποπτεία, τραπεζική εποπτεία, ενώ δεν τα κατάφεραν και τόσο καλά στη δική τους εποπτεία. Εμείς δεν ζητάμε βοήθεια. Θέλουμε να είμαστε παρατηρητές στο σύστημα και δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τις αποφάσεις που λαμβάνουν αυτοί οι οποίοι δεν μπορούσαν καν να υποπτεύσουν τις δικές τους τράπεζες. <clears throat> και αυτό το λέμε. Όχι γιατί θέλουμε να, να, να ξεφύγουμε από το σύστημα. Θέλουμε να συμμετέχουμε στο σύστημα επίση όρις. Αλλά θέλουμε επίση να κατανοήσετε πω εμεί μπήκαμε σε αυτή την ένωση για να συνεργαστούμε με τις υπόλοιπες χώρες, να οικοδομήσουμε την ενιαία αγορά και δεν μπορεί να υπάρχει μια τέτοια κατάσταση όπου στην ενιαία αγορά ε, υπάρχουν ε, άνθρωποι που έχουν δικαιώματα και άλλοι που δεν έχουν. Με εντυπωσιάζει λοιπόν η σημερινή συζήτηση. Ε, με εντυπωσιάζει γιατί οι συνάδελφοι που ήταν πολύ σταθερή στην υπεράσπιση της ενιαίας αγοράς και αυτό είναι πολύ σωστό γιατί όντως φτιάχνοντας την ενιαία τραπεζική αγορά το τελευταίο που θέλουμε να κάνουμε είναι να διαλύσουμε την ενιαία αγορά. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Λάγκεν. Ο κύριος Λάγκεν είπε έχουμε εποπτεία και η εποπτεία μας δουλεύει. Έχουμε ακριβώς και υποδειγματική εποπτεία. Εφόσον λοιπόν έχουμε εποπτεία που λειτουργεί, μπορούμε να συγχωνεύσουμε την τεχνογνωσία που έχουμε, να συνδυάσουμε τον κόσμο, αλλά δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα εκτελώ νέο σύστημα και να ε, εξαφανίσουμε, να διαλύσουμε το παλιό. Και όσον αφορά αυτήν την ιδέα του ελέγχου των μικρότερων τραπεζών από το, ένα κεντρικό επόπτη, Μα Λυπάμαι, μα ένα κεντρικό υποπτικό σώμα θα είναι πολύ απομακρυσμένο από την τοπική αγορά των μικρών τραπεζών. Θα καταθέσω λοιπόν τροπολογίες και ε, θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση για αυτά τα θέματα. Θα πρέπει δηλαδή να αποφασίσουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της ε, χρήση του μηχανισμού σταθερότητας στην Ευρώπη. Νομίζω πω αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και σας ευχαριστώ. Ε. Εγώ σας ευχαριστώ. Η κυρία Γκουλάρα τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω να πω δύο-τρία ψηλοπράγματα. Πρώτον, θα δουλέψουμε στη συνέχεια του πακέτου εποπτείας για το οποίο είχαμε συνεργαστεί σωστά και μέσα στο ίδιο πνεύμα. Δηλαδή, νομίζω ο Φιλίπ Λαμπέρτ το είπε ότι είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζουμε εκ των προτέρων πού ε, βρίσκεται η αλήθεια. Πρέπει να γίνουν επιλογές. Τώρα, για την ε, πτυχή ή 17-27, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να διατηρηθεί και να προστατευτεί η εσωτερική αγορά όσο γίνεται περισσότερο, δίνοντας βεβαίως στην Ευρωζώνη τη δυνατότητα να προχωρήσει. Έχω μόνο ένα θέμα, μια ερώτηση, ουσίας και μια πλαισίου. Καταρχήν θα έλεγα ότι όποια επιλογή και αν κάνουμε, θα πρέπει να είμαστε συνεπείς ε, έχω την εντύπωση ωστόσο ότι όλοι θέλουν τα πλανεκτήματα από όλα τα συστήματα και κανένα από τα μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, είναι σαφές ότι η ΕΚΤ αυτή τη στιγμή είναι ισχυρή, διότι έχει μια αναποστολή, έχει όργανα τα οποία είναι δυνατά και ανεξάρτητα και επειδή δεν υπόκειται στο, στα πολιτικά παιχνίδια Πώς μπορούμε να έχουμε όλα τα ωφέλη της ΕΚΤ έχοντας ένα όργανο το οποίο θα είναι πιο υποχρεωμένο να συνεργάζεται με τους πολιτικούς, την εξαρτησία του οποίου θα είναι ίσως πιο αμφιζητήσιμη κτλ. Εφόσον θέλουμε την ΕΚΤ θα χρησιμοποιήσουμε την ΕΚΤ και να μην ονειρευόμαστε ε, ότι θα είναι κάτι που το οποίο θα είναι τελείως ανεξάρτητο και ταυτόχρονα τελείως υπόλογο ε, στο, στην πολιτική. Τα, δηλαδή να είναι απόλυτα έκτη και απόλυτα ενιαία αγορά. Ε, το, κάθε σύστημα έχει τα υπέρ και τα κατά του. Και ήδη γίνεται λόγος για τα κατά, για, ε, τον γερμανικό τύπο. Επίσης να πω τι γίνεται με το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό του Συμβουλίου. Ε, το, με το Συμβούλιο του Ιουνίου, με συγχωρείτε. Έπρεπε να φτιαχτεί μια τραπεζική εποπτεία για να μπορέσουμε ακριβώς να ανακεφαλοποιήσουμε τις τράπεζες υπό καλές συνθήκες. Και εδώ, Βέρνερ, όταν λέμε ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, υπάρχουν μικρές τράπεζες που μπορεί να δημιουργήσουν κίνδυνο. Βεβαίως δεν θέλουμε να ελέγξουμε τα πάντα με όλες τις λεπτομέρειες. Το κριτήριο δεν είναι μικρό ή μεγάλο, αλλά ότι στο, σε όλα τα κατημέρια θα πρέπει να ελέγχονται τα ίδια, του ίδιου τύπου ιδρύματα. Είπαμε, ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, πρέπει να ενισχυθεί η εποπτεία γι' αυτό. Ε, ωραία, η Μαριάν ε, το έχει πει ότι ήμασταν ανέκαθεν υπέρ. Εντάξει, πάμε γρήγορα. Και τι θα γίνει άμα δεν πάμε γρήγορα. Ότι δηλαδή όσα είχαμε πει για την ανακεφαλαιοποίηση θα περιμένουν για να τελειώσουμε εμεί τις εργασίες μας. Είναι ένα σημαντικό ερώτημα. Από ό,τι είπε ο Μισελ Μπαρνιέ, επέλεξαν ε, αυτό αυτή τη διαδικασία. Για, τώρα άμα το Συμβούλιο έχει αλλάξει γνώμη, είπε ότι μετά και μετά τα ξεείπε, Εκεί είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Τι θα γίνει για μια χώρα όπως η Ισπανία να αργήσει η διαδικασία, τι θα γίνει για την ε, διαδικασία ΕΣΕΜ. Δίνουμε την εντύπωση σε ότι έχουμε κάποια μέσα τελικά και μέσα σε αυτό το πνεύμα νομίζω θα πρέπει να δουλέψουμε όσο γίνεται πιο ε, γρήγορα και φυσικά καταλαβαίνω το ενδιαφέρον εφόσον τόσοι συνάδελφοι συμμετείχαν στη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Δεν έχουν ζητήσει άλλοι το λόγο και γι' αυτό στρέφομαι στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η συζήτηση που προηγήθηκε ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Αναφερθήκατε εσείς και οι συνάδελφοί σας σε όλα τα θέματα τα οποία θεωρούμε και εμείς σημαντικά. Αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί ε, σε αυτή τη φάση το Συμβούλιο έχει αρχίσει να επεξεργάζεται την πρότασή μας την νομοθετική. Η πρώτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου θα ε, διεξαχθεί αύριο και μεθαύριο. Και αισθανόμεθα, θα έλεγα, ότι υπάρχει πραγματική επιθυμία στο Συμβούλιο οι διαπραγματεύσεις αυτές να προχωρήσουν με αρκετή ταχύτητα. Πάρα πολλά θέματα uh, ECB... E Έχουν τεθεί πολλά θέματα σχετικά με το γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να αναλάβει την εποπτεία του πιστοτικού ευρωπαϊκού χώρου και ίσως και πέραν αυτού. Αυτή είναι επιλογή της συνάντησης κορυφής της ζώνης ευρώ της 29ης Ιουνίου. Εμείς αναλύσαμε με επιμέλεια πιστεύω την επιλογή αυτή και αποφασίσαμε να δώσουμε συνέχεια λοιπόν στην επιλογή αυτή του Συμβουλίου για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Πρώτον, γιατί πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει την δυνατότητα, έχει την εμπειρογνωμοσύνη, έχει την ανεξαρτησία ε, και την εμπιστοσύνη που απαιτείται για να το κάνει αυτό, την αξιοπιστία. Γνωρίζουν, ε, γνωρίζουμε βέβαια ότι υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιες αρνητικές πλευρές. η δυσκολία σαν παράδειγμα του να έχουν τα ίδια δικαιώματα στο Εποπτικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των χωρών που συμμετέχουν αλλά και των χωρών που συνεργάζονται. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που μας απασχολούν. Οφείλουμε όμως να αναγνωρίσουμε ότι θα υπήρχαν αρνητικές επιλογές ακόμα και αν ακολουθούσαμε διαφορετικούς κανόνες. Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα νέο σώμα, εντελώς καινοτόμο, εκτός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και δεν είμαστε πεπισμένοι ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πραγματική ενίσχυση της ουσιαστικής εποπτείας των ε, ε, πιστοτικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από τα θετικά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ότι δεν έχει νομικούς περιορισμούς, κάποιους νομικούς περιορισμούς που έχουμε εμείς επανειλημμένα συζητήσει σχετικά με την υπόθεση, με την ομολογία Μαρώνη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να ασκήσει την εποπτεία με διακριτική ευχέρεια χωρίς να περιορίζεται από την ομολογία αυτή, κάτι το οποίο θα ήταν πολύ πιο δύσκολο για ένα νέο σώμα ή για το EBA, την Ευρωπαϊκή Πιστοτική Αρχή, Τραπεζική Αρχή. Λοιπόν, όπως είπε και η κυρία Γκουλάρ, ε, υπάρχουν αρνητικές πλευρές, αλλά έτσι κι αλλιώς θα υπήρχαν αρνητικές πλευρές, ακόμα κι αν κάναμε μια διαφορετική πρόταση. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο προσπαθήσαμε και αποφασίσαμε να συγκλίνουμε ε, προς την κατεύθυνση αυτή το έχει πει ο κύριος Μισελ Μπαρνιέ, ο αρμόδιος επίτροπος. Πάνω σε ένα τόσο σημαντικό θέμα, αυτό το οποίο απαιτείται είναι να δημιουργηθεί σύγκληση ανάμεσα στα θεσμικά όργανα το ταχύτερο δυνατόν. Δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος να δράσουμε με διαφορετικό τρόπο από αυτόν τον οποίο πρότεινε η συνάντηση κορυφής της Ευρωζώνης. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή σύγκληση ανάμεσα στα όργανα τα θεσμικά και ελπίζω αυτό να το κάνουμε το ταχύτερο δυνατόν και με το Συμβούλιο και με το Κοινοβούλιο. Ένα αρνητικό σημείο της χρήσης του 126, του άρθρου 126 της συνθήκης είναι ότι δεν είμαστε στη διαδικασία συναπόφασης. Η Επιτροπή όμως διευκρίνησε ότι εμείς πιστεύουμε ότι οι προτάσεις αυτές αποτελούν ένα πακέτο και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη και των τριών οργάνων για τις δύο αυτές προτάσεις. Αυτό είναι το πνεύμα με το οποίο θα ξεκινήσουμε τις συζητήσεις. Τέλος, για το χρονοδιάγραμμα κατανοώ τους ε, συναδέλφους σας οι οποίοι ζήτησαν να υπάρξει προσοχή, επιφυλακτικότητα, να μην βιαστούμε εν πάση περιπτώσει. Αυτό το δέχομαι απολύτως. Ταυτόχρονα έχει δημιουργηθεί μια κάποια όθηση τώρα θα έλεγα σε σχέση με την πολιτική αυτή διαδικασία και αυτή την όθηση προς τα εμπρός ε, δεν θα ήταν καλό να την απολέσουμε. Θα ήταν πράγματι λυπηρό εάν παραμείνουμε σε επίπεδο απλών συζητήσεων ε, για τα δύο αυτά τα θέματα και το 2013. Αυτό θα το δουν οι αγορές με πολύ κακό μάτι. Αυτό δεν θα αρέσει ούτε στους πολίτες και η διεθνής μας θέση δεν θα τονιστεί. Να μην ξεχνάμε λοιπόν ότι οι δύο αυτές νομοθετικές προτάσεις στην ουσία είναι μια απόπειρα να δώσουν ένα τμήμα της απάντησης στην κρίση από πλευράς της Ευρωζώνης και γι' αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθούν και να εφαρμοστούν το ταχύτερο δυνατόν. Θεωρώ ότι το χρονοδιάγραμμα μέχρι τον μήνα Δεκέμβριο είναι αρκετά φιλόδοξο. Από την άλλη όμως, λαμβανωμένη της δικής σας εμπειρίας, λαμβανομένη της ε, πείρας που έχει σωρεύσει και το Συμβούλιο, νομίζω ότι μπορούμε τον Δεκέμβριο να καταλήξουμε σε μια πρώτη ε, κοινή θέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απολύτως διαθέσιμη να συνδράμει και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε, ό,τι τεχνικό, σε όποιο τεχνικό επίπεδο το επιθυμούν. Ε, επιστρέφουμε στους εισηγητές μας. Α, ο κύριος Γκοζές. Κύριε Πρόεδρε, να επανέλθω στο θέμα του χρονοδιαγράμματος πριν δώσετε το λόγο στους εισηγητές και αφού ακούσαμε την Επιτροπή. Είναι σαφές ότι πρέπει να πάμε γρήγορα λόγω της κρίσης, πρέπει να προτείνουμε λύσεις, πρέπει ο μηχανισμός χρηματοδότησης να λειτουργήσει. Από την άλλη ε, δεν μπορούμε να μην ακούνε, ακούμε αυτά που λένε οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Άκουσα ότι η Γαλλία και η Γερμανία συμφωνούσαν λέγοντας ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος. Οι χώρες αποφασίζουν βέβαια και κάνουν ό,τι επιθυμούν αλλά για να είμαστε σοβαροί εμείς δεν μπορούμε να ε, λειτουργήσουμε μέσα σε πάρα πολύ στενές χρονικές προθεσμίες. Από πλευράς λοιπόν ε, του ΕΛΚ εμείς ζητάμε να παραταθεί η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών και των εκθέσεων βέβαια και νομίζω ότι αν ε, ξεφύγουμε έστω και λίγες εβδομάδες χρονικά πάλι θα τελειώσουμε πριν από το Συμβούλιο, στοιχηματίζω. Θα ήθελα επίσης ότι ξαφνικά η Επιτροπή μας θυμίζει την απόφαση του δικαστηρίου Μωρώνη. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχει μια Ευρώπη η οποία κινείται προς τα εμπρός και υπάρχει και μια απόφαση τεσσαρακονταετίας η οποία μας, ε, μας λειτουργεί σαν τροχοπέδι. Κοιτάξτε, νόμιζα ότι το είχαμε θάψει αυτό όταν μιλήσαμε για πρώτη φορά ε, το θέμα της εποπτείας θα πρέπει ο νομοθέτης εν πάση περιπτώσει, έτσι έμαθα εγώ όταν σπούδαζα νομικά, ότι ο νομοθέτης είναι αυτός ο οποίος μπορεί ε, να κυριαρχεί επί της νομολογίας και δεν θα πρέπει οι ανόητες αυτές τις παλιές αποφάσεις να μας δεσμεύουν. Σας ευχαριστώ. Α, η κυρία Γκουλά. Όχι, απλώς ήθελα να ρωτήσω κάτι το Ζαν Πολ. Βεβαίως χρειαζόμαστε χρόνο για να λειτουργήσουμε σωστά, αλλά ε, πώς σκέφτεται το χρονοδιάγραμμα. Λίγες εβδομάδες τι σημαίνει αυτό, πώς μεταφράζεται στο χρονοδιάγραμμα. Και επίσης, όντως πιστεύω ότι έχει τη στρατηγική του σημασία το Κοινοβούλιο να δείξει ότι μπορεί να εργάζεται και γρήγορα. Και πριν το Συμβούλιο δυνατόν να ολοκληρώσουμε. Δεν υπάρχει κανένα λόγος να χρονοτριβούμε. Μικρή προθεσμία εντάξει, αλλά μην το στείλουμε και στις καλένδες. Μα νομίζω ότι η γραμματεία, λέει ο κύριος Γκοζές, έχει κοιτάξει τις τεχνικές δυνατότητες. Να έχουμε αρκετό χρόνο για να εργαστούμε σωστά, αλλά και να φτάσουμε ε, εγκαίρως και πριν το Συμβούλιο. Νομίζω ο Πρόεδρος μπορεί ε, να τα ανακοινώσει. Μου έδειξαν τις ημερομηνίε, αλλά δεν είναι δική μου δουλειά, τη κοινοποιήσω. Και οι δύο εισηγητές συμφωνούν στις 22 Οκτωβρίου να ζητήσουμε το σχέδιο της έκθεσής τους, ενώ η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών να λήγει στις 26 Οκτωβρίου. Έρχομαι ξανά στους ηγητές, κυρία Τάισεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πραγματικά ε, με εντυπωσίασε πολύ ε, το εύστοχο των παρατηρήσεων όλων των ομιλητών. Είναι πάρα πολύ καλή συζήτηση, πάρα πολύ επίκαιρη και το θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Το αντιληφθήκαμε όλοι. Άκουσα φωνές υπέρ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κατά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Ε, είναι ένα δίλημα αυτό. Άκουσα πολλά επιχειρήματα και έχω και μεγάλη κατανόηση για αυτά, αλλά όλα συμφωνούν με τις ίδιες ανησυχίες και τα μελήματα που σας σκιαγράφησα και εγώ στην αρχή. Τι πρέπει να φροντίσουμε. Όλα τα επιχειρήματα που άκουσα προς τη μία την άλλη κατεύθυνση εκινούν από την ίδια αυτή ανησυχία. Λοιπόν, τα μελήματά μας σε αυτά τα θέματα που μας απασχολούν είναι κοινά και κάπου ελπίζω να καταλήξουμε και από κοινού. Γνωρίζουμε ότι εργαζόμενοι τώρα επί της προτάσεως αυτής θα καταλήξουμε σε ένα μηχανισμό γύρω από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό έχει αρκετούς περιορισμούς. Ε, εντάξει, η νομολογία την αφήσουμε στην άκρη, αλλά υπάρχει συνθήκη και το κανονισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό δεν μπορούμε να τα παρακάμψουμε. Ε, υπάρχει ένας, ε, ένα κανονιστικό πλαίσιο που κάπως μας περιορίζει. Αλλά τι να κάνουμε. Από την άλλη όμως, και σωστά ακούστηκε, υπάρχει μία όθηση προς τα εμπρός, μια ορμή, κάτι γίνεται, ένα κλίμα ότι επιτέλους κάτι να γίνει, αυτό που ζητάμε εδώ και χρόνια, μια διετία τουλάχιστον, μια ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία. Έχουμε την ευκαιρία να το επηρεάσουμε ή μπορούμε να το αφήσουμε να πάει χαμένο, να αρχίσουμε από την αρχή να τα απορρίπτουμε σε λίβδιν ε, και να είμαστε απ' έξω. Όχι. Ε, και κοιτάξτε, δεν εργαζόμαστε και στο κενό, το είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Υπάρχει πολιτική συμφωνία που έγινε σε επίπεδο ε, αρχηγών κρατών κυβερνήσεων της Ευρωζώνης. 17 ηγέτες συμφώνησαν εκεί. Δεν είναι και αυτό ασήμαντο. Ούτε μπορούμε να πούμε ότι είναι ε, ε εντάξει, ένα δευτερεύον περιστατικό. Ήταν σημαντική αυτή η ανακοίνωση. Ε, έχει έρθει πρώτα σε Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τώρα είναι η σειρά μας να διαμορφώσουμε τη θέση μας. Εγώ λοιπόν την προτείνω, Πρόεδρε να δούμε ποια είναι τα θέματα που μας προβληματίζουν και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε, πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε τις προτάσεις που έχουμε επιτάπητος και όσο γίνεται να παραμείνουμε ενωμένοι, συμπαγείς και 27, να μην υπάρχει εκεί μια διαίρεση 17 απέναντι στους 27. Έχουμε μια εσωτερική αγορά, θέλουμε ολοκλήρωση της Ένωσης, όχι διάλυση της. Αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους τους συναδέλφους. Στην πρόταση λοιπόν που έχουμε ενώπιό μας θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί αυτό να βελτιωθεί. Πώς μπορούμε να φροντίσουμε να υπάρχει και ελκυστικότητα για κράτη-μέλη που δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης δεν λέω να είναι μεγαλύτερη ελκυστικότητα, αλλά υπάρχει καν ελκυστικότητα, γιατί δεν είναι καθόλου ε, ελκυστική. Τώρα είναι στη διακριτική ευκαιρία του καθενός, εκτός από τα όργανα εκείνα που έχουν την αρμοδιότητα να το προσδιορίσει αυτό. Μπορούμε να δούμε τις ε, προϋποθέσεις για μια στενότερη συνεργασία και να τις βελτιώσουμε υπέρ των κρατών που θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το σύστημα. Επίσης να δούμε και το καθεστώς των χωρών που δεν είναι στην Ευρωζώνη και πώς μπορούν να συμμετέχουν στο Εποπτικό Συμβούλιο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με αυτό το καθεστώς, πώς μπορούν να συμμετέχουν αυτές οι χώρες και επίσης ε, τι κύρος θα έχει και τι ευθύνη ε, και για ποια πράγματα θα αποφέρεται αυτό το Εποπτικό Συμβούλιο. και πώς θα γίνει αυτό στο εσωτερικό μιας Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που καλός ή κακός ή δυστυχώς, δεν ξέρω, διαπίστωση είναι, ε, έχει ένα όργανο λήψη αποφάσεων μεταβατικό αφού υπάρχει εξαίρεση για κάποια κράτη-μέλη. Λοιπόν, πώς μπορούμε, αν μπορούμε να ενισχύσουμε το ρόλο αυτού του συμβαλίου και πώς θα γίνει αυτό. Έχω χώρες της αλλά και χώρες που δεν συμμετέχουν στην Ευρωζώνη. Να δούμε τι μπορεί να γίνει νομικά και τι επιτρέπει η συνθήκη, το κείμενο ε, νομοθετικό πλαίσιο. Και τώρα για τις τράπεζες. Ο κύριος Κλίντς νομίζω το είπε για τις ασφάλειες. Μα είπαμε αν είναι νομική βάση 127.6 είναι έξω ασφαλιστικές εταιρείες, οργανισμοί, οτιδήποτε επιχειρήσεις ασφαλιστικές, είναι μόνο οι τράπεζες. Πρέπει να το γνωρίζουμε, το ορίζει αυτό η συνθήκη, δεν μπορούμε να βάλουμε τις ασφάλειες. Είναι σαφέστατο άμα πάει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι ένας περιορισμός, μπορεί να μας αρέσει ή όχι, αν μπούμε στην ΕΚ, την έξω οι ασφάλειες. Τώρα, τράπεζες είπαμε. Ναι, αλλά ποιες τράπεζες τώρα. Εκεί ακούσαμε πολλά. Δεν θέλουν όλοι να μπαίνουν άμεσα σε αυτή την εποπτεία όλες οι τράπεζες με ένα κεντρικό επόπτη. Αφήστε που κάτι τέτοιο μπορεί να μην είναι και εφαρμόσιμο στην πράξη. Λοιπόν, ποιες τράπεζες θα μπουν στην άμεση εποπτεία, ποιες τράπεζες παραμένουν στην εθνική εποπτεία και να φροντίσουμε να υπάρχει ένα, σημαντικό, ένα ενιαίο μάλλον σύστημα ε, εθνικών εποπτών αυτό μπορούμε να το δούμε με κάποιο τρόπο υπολογισμού. Matrix, που ακούσαμε και στις 3 Σεπτεμβρίου ότι μπορεί να γίνει αυτό στην ακρόαση, ε, προς τα εκεί να κινηθούμε. Τώρα, ποια θα είναι τα καθήκοντα, ποιος αναλαμβάνει ποια ευθύνη και ποια υποχρέωση, τι γίνεται με τους εθνικούς επόπτες, τι γίνεται με τον Ευρωπαίο, τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, EBA. Όλα αυτά επίσης να τα κοιτάξουμε και να δούμε, έχουμε κάποιο περιθώριο λιγμών. Κάτι άλλο που έχει σημασία και ερχόμαστε εδώ στη λογοδοσία. Αν παραμείνει αυτή η δομή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ας κάνουμε αυτή την υπόθεση εργασίας, τότε εμείς έχουμε μικρότερο λόγο μεν για τα όσα συμβαίνουν εκεί. Αλλά ε, όσο αυξάνεται η ανεξαρτησία μαζί με τις εξουσίες ε, του οργάνου, θα πρέπει να συμμετέχει και το Κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε όλα στο εποπτικό συμβούλιο και τα των τραπεζών και τα υπόλοιπα. Μου φαίνεται πάρα πολύ ευρύ εντολή αυτή. Και στον κανονισμό θα πρέπει να ρυθμίζονται πολύ περισσότερα και να μην είναι στη διακριτική ευκαιρία του εποπτικού συμβουλίου για το πώς θα λαμβάνουν αποφάσεις, πώς θα... όπως και να ψηφίζουν. Για την ανεξαρτησία το συνικό τείχος ή όποιο άλλο τείχος ανάμεσα στα εποπτικά και τα νομισματικά. Ακριβώς να δούμε τι καθεστώς μπορούμε να δώσουμε στο εποπτικό συμβούλιο. Ποια είναι η σχέση του με τα όργανα που λαμβάνουν αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γιατί εκεί μπορεί να χρειάζεται κάποια ρύθμιση και μπορούμε να το ενισχύσουμε. Και έρχομαι στη δημοκρατική λογοδοσία, όσο ε, κατοχυρώνεται αυτή η αρχιτεκτονική στη συνθήκη, τόσο πώς να το πω, ε, περισσότερες αξιώσεις και, ε, ε, μπορεί να έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για διαφάνεια και συμμετοχή. Αυτό μπορούμε να το ενισχύσουμε, χωρίς να δημιουργήσουμε ένα ιδανικό κόσμο, αλλά τον έλεγχο βεβαίως μπορούμε να τον ισχύσουμε. Ε, έγινε μεγάλος λόγος για το ποια θα είναι η στέγη της ε, εποπτικής αυτής αρχής, η EBA, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ε, κάποια στιγμή θα απαντηθεί και αυτό, δεν ξέρω. Και τέλος, Πρόεδρε, νομική συμβολή θα μπορούσαμε να ζητήσουμε ε, για το μέχρι πού μπορούμε να τροποποιήσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να συμπεριλάβουμε τα μελήματα όλων των συναδέλφων. Αυτές είναι οι προτάσεις μου. Περιμένετε σε λίγες εβδομάδες να φέρω ένα σχέδιο έκθεσης. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθώ, εάν συμφωνείτε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε μέσα σε λίγες εβδομάδες Ε, εκτός να πούμε ότι το απορρίπτουμε σε Λίβδιν και ζητούμε άλλη πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι. Ε, το θέμα, ε, και μετά θα έχουμε απέναντι το Κοφίν και τους άλλους, πρώτα να κοιτάξουμε τι μπορούμε να κάνουμε με την πρόταση που έχουμε, την παρούσα και αλλιώς να κοιτάξουμε τι άλλες δυνατότητες υπάρχουν. Το είπε και η Σιλβί Γκουλάρ. Δεν δουλεύουμε στο κενό. υπάρχει και επίγουσα κατάσταση. Δεν είναι μόνο οι μπάνκια στην Ισπανία. Έχουμε μια κρίση, ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει το παραμικρό και ε, ακόμα ψάχνουμε <laughs> την εμπιστοσύνη. Είπαμε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη με την πρόταση αυτή και αν το απορρίψουμε από την πρώτη μέρα ότι τι είναι αυτά τα πράγματα που μας προτείνεται ποτέ των ποτών δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε φέρτε άλλη πρόταση ε, τότε χάος δημιουργούμε και θα έχουμε και χαόδεις αντιδράσεις και ε, μπορούν να το εκμεταλλευτούν αυτό και οι αγορέ. Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι του συναδέλφου. Ήταν πάρα πολύ καλή και πολύτιμη η συζήτηση και θα με βοηθήσει οπωσδήποτε για να κάνω εγώ τη δουλειά μου για τον κανονισμό αυτό όσο γίνεται καλύτερη. Θα σας φέρω ε, την πρόταση, θα, θα συγγράψω όλα αυτά που προτείνατε εσείς. Εξάλλου αυτός είναι ο λόγος του εισηγητή. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Γκίγκολτ. Θα ήθελα απλά να κάνω κάποια σύντομα σχόλια μετά από τη συζήτηση. Για τα βασικά κριτήρια για το τι θέλουμε να επιτύχουμε, άκουσα πολλά κοινά, κοινές επιθυμίες. Ενίσχυση ε, ε, η, διατήρηση όσο γίνεται της συνοχής για τον κανονισμό της ενίας αγοράς, αποτελεσματικότητα του συστήματος, ε, χωρίς να δημιουργούνται επιπλέον προβλήματα. Αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να δίνονται σαφείς εξηγήσεις για τους ομίλους και φυσικά το θέμα της δημοκρατικής λογοδοσίας. Εγώ νομίζω πως εδώ λοιπόν κινούμαστε όχι προς ένα πολύ σοβαρό πολιτικό πρόβλημα, απλώς αγγίζουμε κάποια όρια της νομικής πρότασης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει σοβαρά να λάβουμε υπόψη. Και μπορούμε τώρα να ακολουθήσουμε δύο δρόμους. Να πούμε δηλαδή βασικά ότι αυτά είναι τα προβλήματα τα νομικά, τα αφήνουμε στην άκρη, στο πλαίσιο της ε, τωρινής πρότασης όμως. Και μετά πρέπει να εξολογήσουμε πόσο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και αν αυτό δεν αρκεί ε, με βάση τα πολιτικά κριτήρια, τότε βέβαια θα πρέπει σαφώς να σκεφτούμε κατά πόσο θα παραδοθούμε με τον νόμο ή κατά πόσο θα πρέπει να ισχύουν πολιτικά κριτήρια για να μπορούμε να αλλάξουμε την νομοθεσία. Αυτό είναι ο ρόλος μας και εδώ πρέπει να προσέξουμε πάρα, πάρα πολύ, αλλά φυσικά δεν λειτουργούμε εν κενό και πρέπει να είμαστε σε θέση να φτιάξουμε κάτι το οποίο να μπορεί να δώσει την ισχυρή τραπεζική εποπτεία που χρειάζεται η Ένωση. Και ε, ε, αυτές θα είναι οι βασικές ε, διαπραγματεύσεις. Απλώς θέλω να κάνω μια δημόσια πρόσκληση σε μια συνάντηση με, νομικού νομικούς αύριο το πρωί για να συζητήσουμε αυτούς τους περιορισμούς της υπόθεσης Μαρόνι γιατί υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το τι ακριβώς σημαίνει αυτή η υπόθεση Μαρόνι. Και αυτό είναι υποσυζήτηση και θέλω να αναφέρω ε, μόλις δύο ε, παρατηρήσεις. Η παλαιά απόφαση τη Μαρόνη ήταν ότι ο προκάτοχος της Κομισιόν στην ουσία ανέθετε καθήκοντα σε ένα τελείω μη δημοκρατικό χώρο. Εδώ όμως μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό, ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να θέτουν στην έκτη κάποιες αρμοδιότητες, κάτι πολύ διαφορετικό. Στην υπόθεση Μαρών, λοιπόν, όπως, όπως ανέφερε ο συνάδελφος Ζαν Πόλε, φτιάχτηκε ένας ολόκληρος πύργος της ε, Βαβυλώνας και όλοι φοβόντουσαν της Βαβέλ, συγγνώμη, και όλοι αναρωτιόνταν ε, τι νόημα είχε αυτό και θέλω να το συζητήσω με την Κομισιόν κατά πόσο δηλαδή η υπόθεση Μαρών είναι μια βάση όπου δεν μπορεί κανείς εύκολα να μετακινήσει και να μεταβιβάσει τόσο ευρία καθήκοντα στην ΕΚΤ. Και το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και στο μέλλον να το συζητήσουμε. Δεν μπορούμε να δεχτούμε, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι στο πλαίσιο της ΣΕΚΤ θα έχουμε μέλη με διαφορετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις. Θα πρέπει να είναι κοινά και αυτή είναι μια πολύ βασική αρχή τα όσα είπε ο, ο, συνάδελφος από την Πολωνία είναι απόλυτα κατανοητά και Άκουσα μάλιστα και δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει ότι μάλιστα το πρώτο σχέδιο της πρότασης της Κομισιόν το συμπεριλάμβανε αυτό και αργότερα ε, έγιναν κάποιες εσωτερικές συζητήσεις με τη δική τους νομική υπηρεσία που είπε ότι κάτι τέτοιο δεν θα είναι δυνατόν. Υπάρχουν δηλαδή πολλά νομικά θέματα για το τι μπορεί να κάνει κανείς μέσα στην ΕΚΤ σε σχέση με αυτό που είπε η Μαριάν Τάισεν και θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα ελέγξουμε πολύ πολύ προσεκτικά και αν δεν μπορούμε να επιτύχουμε τα κριτήρια κοινή αγοράς, αποτελεσματική δομή ε, και δημοκρατική λογοδεσία στο πλαίσιο της ΕΚΤ σε αρκετά ευρύ θα πρέπει να έχουμε το θάρρος και να πούμε ότι τότε χρειαζόμαστε ένα άλλο θεσμό στον οποίο θα συμβάλλει η έκτη με την εμπειρογνωμοσύνη της. Και εκεί υπάρχουν άλλα νομικά θέματα πάλι. Γι' αυτό αν θέλουν αύριο στις 8 να έρθουν οι συνάδελφοι, ευχαρίστως. Τώρα είναι Πάζη που δούλεψε για λογαριασμό μου στη διάρκεια του καλοκαιριού για μένα και για τη συνάδελφο Φρανσίσκα Μπράντνερ. Ε, και γι' αυτό πρέπει να πούμε ότι δεν χρειάζεται επιβεβαίωση του και του Συμβουλίου ότι είμαστε σε συναπόφαση εδώ, γιατί απλούστατα ως Κοινοβούλιο μπορούμε να το θεωρήσουμε όπως ε, ψηφίσαμε στο ψήφισμά μας και σύμφωνα με την ομοφωνία υπό το άρθρο 126.7 ορισμένες χώρες ποτέ δεν πρόκειται να συμφωνήσουν για το 126.7 εάν δεν υπάρχουν δυνατότητες αλλαγής του κανονισμού για την ε, EBA. Βασικά η δική μου πρόταση είναι να επηρεάσουμε ολόκληρο το πακέτο γιατί ορισμένες χώρες ποτέ δεν πρόκειται να υποχωρήσουν χωρίς αλλαγές ε, υπό το άρθρο 126.7 της ΕΜΠΑ δεν πρέπει να ανησυχεί και τόσο πολύ. Αλλά φυσικά η διασύνδεση ανάμεσα στις δύο εκθέσεις σημαίνει επίσης πως εμείς ως ομάδα πρέπει να συνεργαστούμε ανάμεσα στους σκεώδεις των δύο εκθέσεων για να βρούμε μια κοινή θέση. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να τοποθετηθούν πρώτα τα δικά μας πολιτικά κριτήρια και, και το ποιο δρόμο θα ακολουθήσουμε. Ή διαφορετικά θα έχουμε πρόβλημα να βρούμε κοινή βάση. Το χρονοδιάγραμμα είναι κάπως πιο χαλαρό τώρα, αλλά όχι υπερβολικά χαλαρό. Και είναι αυτό μια καλή βάση ώστε να συμπεριφερθούμε υπεύθυνα στη διαδικασία με το Συμβούλιο και εδώ στο ε, Κοινοβούλιο ώστε να επιτύχουμε την πρόοδο που απαιτεί η κρίση του ευρώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Να σας θυμίσω άλλη μια φορά ότι η εξέταση του σχεδίου έκθεσης προβλέπεται για τις 22 Οκτωβρίου και για τις δύο εκθέσεις. <coughs> Και ότι... Ναι, 22 Οκτωβρίου, 22. 22 Οκτωβρίου και η προθεσμία υποβολής τροπολογιών 26 Οκτωβρίου. Τέσσερι μέρες. Να θυμίσω για την έκτατη συνεδρίαση της Επιτροπής ε, την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου από τις 9 μέχρι τις 1. Ακρόαση σε σχέση με την Τραπεζική Ένωση και την διαχείριση της κρίσης. Τέλος της συνεδρίασης.